Good morning, ladies and gentlemen. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. I'm Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω όλους εδώ, παρόντες μετά ε, τις στενές διακοπές. Ελπίζω να περάσετε καλά στις διακοπές σας. Είμαστε έτοιμοι να στρωθούμε στη δουλειά, στη νέα περίοδο που αρχίζει. Καλώς ορίσατε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αρχίζουμε με την έγκριση μερίσιας διάταξης. Ο κ. Βανίστερο έχει κάτι να προτείνει για την ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ πολύ για τα εναρκτήρια λόγια σας. Τώρα έχουμε λίγο προβλήματα να οργανωθούμε, να προσαρμοστούμε. Στην αρχή της ημερήσιας διάταξη είχαμε συμφωνήσει με την Επίτροπο. Πού είναι η Επίτροπος, <laughs> πότε θα έρθει, τι συνέβη, έπαθε τίποτα. Ναι. Ναι. Ήταν σαφής υποτίθεται η ημερήσια διάταξη, το σχέδιο, η ανταλλαγή απόψεων με την Επίτροπο κατά τη διάρκεια του έτους. Ποιο έτους λέει, τώρα λέει ο κ. Βανίστερο. Όχι, όχι. Για όλο το χρόνο είχε δεσμευτεί ότι θα έρχεται. Είχαμε συμφωνήσει ημερομηνίε μεταξύ αυτών και τη σημερινή για το Σεπτέμβριο. Δυστυχώ το πρόγραμμα τη δεν τη επιτρέπει να έρθει στη σημερινή μα συνεδρίαση. Αλλά όπως γνωρίζετε έστειλε μια επιστολή στην Επιτροπή μας, εμένα προσωπικά, την οποία έχετε όλοι λάβει. αναφέρει λίγο πώς έχει η κατάσταση στην προετοιμασία με τις συμφωνίες εταιρική σχέσης και ε, την εξάντε ερεσιμότητα. Δηλώνει προθυμία να έρθει σε επόμενη συνεδρία της Επιτροπής μας. Σήμερα κολλείεται. Είμαι βέβαια ότι θα έρθει, λέει και ο Σβανίστερα, θα έρθει. Και με άλλους επιτρόπους. Α, και άλλη ερώτηση. Έχουμε νέο γενικό διευθυντή. Εκούσαμε τον παλιό. Ο νέος πότε θα έρθει. Ε, αυτό είναι το δεύτερο ερώτημα. Συναντηθήκαμε με τον απερχόμενο, τον απελθόντα και τώρα έχουμε νέο γενικό διευθυντή. Θα τον καλωσορίσουμε πάρα πολύ σύντομα. Η γραμματεία είναι σε επαφή με τις υπηρεσίες ε, του Γενικού Διευθυντή με τη Γενική Διεύθυνση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πολύ γρήγορα θα το δούμε ίσως και την επόμενη φορά. Δεν το γνωρίζω αυτό. Είναι τμήμα και αυτό τη ημερήσια διάταξη. με το έχουμε στο πρόγραμμα. Ευχαριστώ. Τίποτα άλλο για την ημερήσια διάταξη. Όχι. Σα ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε να την εγκρίνουμε λοιπόν. Επόμενο θέμα έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της 13ης και 14ης Ιουλίου. Έχετε ε, στη διάθεσή σας online ε, το σχέδιο των πρακτικών. Αν τη διαφωνήσει κανείς μέχρι το τέλος της συνεδρίασης θα θεωρηθούν εγκεκριμένα τα πρακτικά. Ωραία. Το επόμενο θέμα στη μέση διάταξή μας είναι η έγκριση του σχεδίου χρόνου διαγράμματος των συνεδριάσεων της Επιτροπής μας Ρέτζη για το 2017 οι αρμόδιες υπηρεσίες ε, για το σχεδιασμό των συνεδριάσεων μας και των αντιπροσωπιών ε, και που ασχολούνται με τα θέματα των αιθουσών και της ερμηνείας έχουν καταθέσει ένα χρονοδιάγραμμα για το 2017. Δεν θα μπορώ να σας περιγράψω πόσο δύσκολο είναι αυτό για όλες τις επιτροπές. Ε, βγήκε λοιπόν αυτή η πρόταση από τις υπηρεσίες. Παρακαλώ να την εξετάσετε πάρα πολύ προσεκτικά διότι έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Δεν έχουμε τόσο πολλές πέμπτες απόγευμα, αλλά έχουμε Δευτέρες απόγευμα. Οπότε, σας παρακαλώ, διαβάστε προσεκτικά. Μπορούμε να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε ορισμένε ημερομηνίε, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι θα μπορέσουμε να τα αλλάξουμε όλα από το προτινόμενο αυτό χρονοδιάγραμμα. Μπορούμε να το εγκρίνουμε ή δεν ξέρω, έχετε σχόλια, προτάσεις, θέλει κανείς να πει τίποτα. Όχι. Ας πούμε λοιπόν ότι το εγκρίνουμε και θα προσπαθήσουμε να οργανωθούμε ως προς τα ταξίδια μας. Ευχαριστώ πολύ. Εγκρίνεται το χρονοδιάγραμμα. Ανακοινώσεις της Προέδρου. Δεν έχω τίποτα, απλώς να σας καλωσορίσω και να σας ευχηθώ ε, καλή συνεργασία και γόνιμη κατά τη διάρκεια των επομένων ε, μηνών μέχρι το τέλος του έτους. Είμαι σίγουρη ότι η Επιτροπή Ρέτζι θα συνεχίσει το έργο που παραδοσιακά κάνει και σε μια πολύ καλή και επικοδομητική ατμόσφαιρα. Καλή μας δουλειά λοιπόν μέχρι το τέλος του έτους. Και τώρα θα περάσουμε στις ψηφοφορίες. I'm sorry. We should you can perhaps change the order or ask them if they agree to that. do we have somebody from ECR group? Από την ECR, κανείς. Ο κύριος Πορέμπα έχει κολλήσει σε κάποιο μποτιλιάρισμα και απουσιάζει. Maybe we can change the order. Δεν ξέρω, θέλετε να αλλάξουμε τη σειρά ε, της ψηφοφορίας. Ο κύριος Βον παρευρίσκεται, μάλιστα. Ο κύριος Πορέμπ απουσιάζει. To Δεν θέλετε να αλλάξει η σειρά. Να περάσουμε στην έκθεση του κυρίου Βον. Να ψηφίσουμε. with... We vote with the, the report. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε την έκθεση του κυρίου Πορέμπα. Μέτρα κατοχήριου τη ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο. Είναι ο κανονισμός 994 το 2010. This is the first, what we vote. Αυτό είναι το πρώτο που θα ψηφίσουμε. The, we begin... Ας αρχίσουμε λοιπόν με την Τροπολογία 113. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 114. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 115. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Την τροπολογία 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ. Τροπολογία 116. Υπέρ. Α, καταπίπτει, με συγχωρείτε. Συμβιβαστική τροπολογία 10, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα της συμβαστικής 10, υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Δεύτερο τμήμα της συμβαστικής τροπολογίας 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. περνάμε στην τροπολογία 121. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 127. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 16 καταπίπτει. Περνάμε στην 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 129. Υπέρ. Α, καταπίπτει. Μάλιστα. Συμβιβαστική 14 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 131. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 132. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 134. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 135 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 136 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 137 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 138 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 139 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 140 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 141 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 142 υπέρ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 143. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 144. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 26. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Με συγχωρείτε που ελέγξαμε. 145 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 146 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 148 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 149 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Εκατόν πενήντα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Εκατόν πενήντα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 152. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 153 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 154 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 155 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 157. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 158. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 159. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 160. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 161 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 30 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Όχι, εγκρίνεται, με συγχωρείτε. 162 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 163 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 31 Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 164. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 165. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 166. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 167 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 33 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 34 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 168 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 35 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 171. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 172. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 173. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 174 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 175 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 176 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 36 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική μάλλον τροπολογία 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ Α, με συγχωρείτε. Είμαστε στην τροπολογία 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 54. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 55. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 56. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 57. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές Με συγχωρείτε. Στον κατάλογό μου δεν το είχα. Ναι, θα επιστρέψουμε στην προφορική τροπολογία. Δικό μου το λάθος. Ο δικός μου κατάλογος είναι λάθος, συγγνώμη. Έχουμε λοιπόν μία προφορική τροπολογία. Είναι κάποιος κατά της προφορικής τροπολογίας. Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν τη συμβαστική τροπολογία 5 μαζί με την προφορική τροπολογία. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 66. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ, κατά, Αποχές. Απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Το πρώτο τμήμα εγκρίθηκε, το δεύτερο απορρίφθηκε. Συμβιβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 83 υπέρ κατά, αποχές, ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 83. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 84. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 86 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 87 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 93 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 94 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 97 υπέρ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 99. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 100. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 101. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 106 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. 107. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 108. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 109. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 110. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 111. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 112 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα όλη τη γνωμοδότηση, την έκθεση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω να έχει έρθει ο κύριος Πορέμπα, αλλά θα έρθει αργότερα. the next, the next vote. Η επόμενη ψηφοφορία τώρα αφορά τον ε, Γενικό Προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οικονομικό έτος 2017 όλα τα τμήματα. Ο κύριος Βον είναι ο εισηγητής μας. Θέλετε κάτι να πείτε. Όχι. Ευχαριστώ. Και... And we begin with the compromise one. Πάμε τώρα στην πρώτη συμβαστική τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και πάμε τώρα στην τροπολογία 5. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 6. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 10. Υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 προφορική τροπολογία έχει ζητηθεί έχετε κάποια ένσταση οπότε Ψηφίζουμε το 15 με την προφορική τροπολογία. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. συμβιβαστική 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 17. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. συμβιβαστική 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 19. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21 έχει αποσυρθεί και πάμε στη συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι εγκρίνεται. Θα κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο για την 27. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα η τελική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Πέρας Εγκρίνεται συγχαρητήρια κύριε Βον. Εγκρίνεται και τώρα συνεχίζουμε με ναι, την έκθεση του κυρίου Ρούβας. Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για το Συντονισμό της Οικονομικής Πολιτικής, εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2016. Κύριε Ρούας, θέλετε το λόγο. Όχι. Ευχαριστώ. Ψηφίζουμε. Ξεκινούμε. Πρώτη τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Compromise one In favor. Against. Abstentions. Adopted. Και η δεύτερη εγκρίνεται. Συγγνώμη, η πρώτη εγκρίνεται. Και άρα θα πάμε στην συμβαστική. Δύο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα γίνει ηλεκτρονικός έλεγχο για τη συμβαστική υπαριθμών 2. The vote is closed. Α, εγκρίνεται. Θα πρέπει, θα πρέπει να τα ξαναδώ τα πράγματα. Θα πρέπει να συγκεντρωθώ περισσότερο σήμερα. Αλλά θα, θα το καταφέρω, θα το καταφέρω. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Οπότε πάμε τώρα στην τροπολογία 8. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5 είναι υπομένη, ποιοι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 28. Υπάρχει μέσω προφορική τροπολογία, ενστάσεις. Όχι, επομένω ψηφίζουμε την 28 με την προφορική τροπολογία. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 13. Όχι, συγγνώμη λέει πρόεδρος, συμβιβαστική 6. Εγκρίνεται. 7. Συμβαστική. Υπέρ κατά αποχές και εγκρίνεται. 52. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 53. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Και το τελική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται η έκθεση και σας ευχαριστώ. Τελειώσαμε με τις ψηφοφορίες. Συνεχίζουμε. Το επόμενο σημείο σήμερα είναι η θέσπιση προγράμματος στήριξη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την περίοδο 17 έως 20. Συνεισηγητέ για την Επιτροπή μας είναι η κυρία Κρέλ και ο κύριος Φανίστελτρο και θα εισηγηθούν επί της νομοθετική προτάσεως για την θέσπιση αυτού του προγράμματος στήριξη. Το άρθρο 175 και το άρθρο 197 είναι οι νομικές βάσεις. Και θα πρέπει να αναθεωρηθεί ο κανονισμός των κοινών διατάξεων. Το βασικό τμήμα καλύπτει για την περίοδο αυτή 142,8 εκατομμύρια. Και αφορά τον ε, προϋπολογισμό τεχνικής αρρωγής από το ε, Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Κοινωνικό Ταμείο. Και ζήτησαν οι συγητές να δούμε εάν γίνεται να γίνει και άλλη μία ανταλλαγή απόψεων στην επόμενη συνεδρίαση και να συζητήσουμε τις τροπολογίες. Συμφωνείτε? Οπότε θα έχουμε και την γνωμοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής που είναι συναρμόδια σύμφωνα με το άρθρο 54 αλλά και από την ε, Επιτροπή Επασχόληση σύμφωνα με το άρθρο 53 συν θα γνωμοδοτήσουν αλλά και η Επιτροπή Πολιτιστική αλλά και η Επιτροπή Αλίας που θα γνωμοδοτήσουν σύμφωνα με το άρθρο 53 του κανονισμού. Το τελευταίο που θα σας αναφέρω είναι το εξής. Να ληφθεί υπόψη ότι αυτό αφορά την συνεργασία με την Επιτροπή Περιφερειών. Σύμφωνα με τα όσα συμβαίνουν το 2014. Οπότε και όταν ολοκληρώσουμε τη δουλειά μας και τη γνώμη της εισηγήτριας Επιτροπής των Περιφερειών Ποιος θα ξεκινήσει, κύριε Φανίστορη ή κύριε Κρέλ. Κύριε Φανίστορη. Σας ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή σας αυτή για το θέμα. Δείχνει ακριβώς που βρισκόμαστε, διότι η παρούσα πρόταση ε, καλύπτει ένα ευρύτατο πεδίο ε, εφαρμογής. Βέβαια, η βασική αρμόδια επιτροπή είναι η δική μας αλλά είναι παλιά ιστορία στο Κοινοβούλιο, ποια επιτροπή θα πάρει τι για τις αρμοδιότητες. Έχουμε μια μέθοδο πάρα πολύ διαφωνή, διαφανή ε, και σε κάθε βήμα καλούμε τους συναδέλφους Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων. Είχαμε και επαφές με τα μέλη της Επιτροπής Προεπολογισμών και άλλες ε, επιτροπές που είναι συναρμόδιες για να κάνουμε κοινέ προτάσεις και να ε, περάσει από τη διαδικασία αυτή η λήψη απόφασης φέτος επιτέλους να τελειώνει. Έχετε δίκιο ε, σε αυτό που λέτε. Έχουμε τις τροπολογίες ε, να τις δούμε. είναι τεχνικό το θέμα βασικά, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, διότι ενισχύει τα κράτη-μέλη και τα ενθαρρύνει να κάνουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις καλύτερα και γρηγορότερα. Αν δούμε χώρες όπως η Ελλάδα, με τέτοια εργαλεία και μέσα είναι πάρα πολύ σημαντικό να σταματήσουμε τα λόγια και να περάσουμε σε έργα. Τι, δεν, βοηθάει. Ε, και κάνεις τη δουλειά και παίρνεις την έξτρα υποστήριξη που υπάρχει ήδη, τεχνική υποστήριξη ε, και με τα κονδύλια τα περιφερειακά και του Ταμείου Στρατηγικής Επένδυσης και ιδιαίτερα με το, το, το, το νέο μέσον. Ε, άρα η διαφάνεια, η συνεργασία, η ανοιχτή προσέγγιση ήταν ο γνώμονας και η στάση και γραμμή που τηρήσαμε τους τελευταίους μήνες. Η κυρία Κρέλ και εγώ και οι υπηρεσίες ε, συζητήσαμε με όλους ε, όσοι εμπλέκονται εδώ. Βεβαίως, η Γενική Διεύθυνση, η Ρέγγιο και η Επίτροπος Ρωτήθηκε, μπορούμε να δαπανίσουμε τα τάδε κονδύλια με το δίνα τρόπο. απάντησε, «Ναι, μάλιστα. Αν δείτε τα στοιχεία και η κυρία Κρέλ και εγώ στις διαπραγματεύσεις για την περίοδο 2014-2020 χαρήκαμε πάρα πολύ που για την τεχνική βοήθεια αυξήθηκε κάπως ο προπολογισμό. Και αν τώρα βγείτε και ρωτήσετε, ε, έχουν δεσμευτεί τα κονδύλια αυτά, έχουν δαπανηθεί, απάντηση όχι. Υπάρχει αυτό το πλεόνασμα, ε, η επιπλέον πρικοδότηση. Ε, και ε, στη θέση αυτή του προϋπολογισμού περίπου έχουν φύγει τα κονδύλια από εμά και έχουν ενταχθεί σε αυτή τη νέα πρόταση με το νέο σχήμα. Τώρα, σήμερα αυτό δεν επηρεάζει αυτές κατά τις δικές μας προτεραιότητες ή την τεχνική βοήθεια. Αυτό είναι κάτι που ζητάμε ξανά και ξανά, πάγιο αίτημα. Δεύτερο, για τις τροπολογίες, αυτές ενισχύουν την πρόταση. Δεν θα είναι κανένα μετέωρο νέο ταμείο που θα άγεται και θα φέρεται. Αν δείτε τη λέει Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αναφορά της, τα δύο τρίτα των συστάσεων αναχώρα έχουν σχέση με τη συνοχή. Ε, ε, καλά, σας δεν χρειάζεται εδώ να σας πείσω στην Επιτροπή ότι ε, τα δικά μας κονδύλια είναι πάρα πολύ σημαντικά για την ανάκαμψη της οικονομίας και για τις μακροχρόνιες αλλαγές. Είναι γνωστά αυτά και βρισκόμαστε στη βάση ενός τριγώνου. Το τρίγωνο έχει τρεις πλευρές ως γνωστό, οπότε είναι και το θέμα της απασχόλησης, της ανάπτυξης, ε, για το περιβάλλον, για τα ε, ε, θέματα ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Με τις τροπολογίες μας λοιπόν τι θέλουμε, να ενισχύσουμε αυτό το ταμείο, να έχει καλύτερη συνάφεια με τη δική μας πολιτική συνοχή και τους στόχους και δεν μπαίνουμε στα χωράφια της ΕΚΟΝ τα οικονομικά, δεν μπαίνουμε σε αλλαγέ, α πούμε, σε τραπεζικά συστήματα και τέτοια. Δεν μα ενδιαφέρουν αυτά. Εμεί δεν είμαστε χρηματοπιστωτική επιτροπή, ούτε τραπεζική επιτροπή εδώ. Έχουμε ε, πάντως αυτό το φάκελο ω ε, καθήλυνα και υιοθετήσαμε αυτή την προσέγγιση. Μάλιστα, τη δουλειά μας την κάναμε νομίζω και θα απευθυνθώ στην κυρία Κρέλ. Δεν ξέρω, τα καλύψαμε όλα σχεδόν τα θέματα, δεν σκέφτομαι τίποτα. Ίσως η κυρία Κρέλ να έχει να πει κάτι παραπάνω. Αν μου επιτρέπει η πρόεδρο να σα δώσω το λόγο. Βεβαίω, Λάμπερτ. Η κυρία Κρέλ έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για την ε, καλή συνεργασία, ιδιαίτερα τον Λάμπερτ και τη Γραμματεία. Στην αρχή υπήρξε κάποια σύγχυση για ε, τις ε, αρμοδιότητες, για το αν αυτό είναι μια ευθεία επίθεση του, κατά του σχεδίου Γιούγκερ, κατά της ε, διαρθρωτικής πολιτικής. Όμως, με, δεύτερη, με τη δεύτερη σκέψη, τρίτη σκέψη, είδαμε ότι είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα, ότι εδώ δεν προσπαθούμε να καταστρέψουμε την πολιτική συνοχής. Και να πω επίσης ότι είχαμε εξαιρετική εμπειρία με την Task Force στην Ελλάδα που έδωσε τη δυνατότητα στην Ελλάδα να ε, απορροφήσει 100% σχεδόν των ε, διαθερωτικών ταμείων και αυτό μέσω της τεχνικής υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θεωρώ λοιπόν πως είναι μια καλή ιδέα τα ε, κονδύλια που υπολείπονται για την τεχνική υποστήριξη να ε, τα αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να τα διαθέσει στις χώρες που τα ζητούν. Ε, είναι προαιρετική ε, αυτή η χρήση. Θα τα ζητούν προαιρετικά. Θα παρέχεται τεχνική στήριξη. Θεωρώ λοιπόν πως είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα και νομίζω εξάλλου ότι στο σχέδιο έκθεσης καθίσταται σαφές ότι κατά κύριο λόγο θα στηρίζονται προγράμματα μεταρρυθμίσεων τα οποία θα ε, έχουν ως στόχο να ε, επιτυγχάνουν την συνοχή. Επίσης ε, δεν πρέπει να δημιουργηθεί προηγούμενο σε σχέση με την ε, χρηματοδότηση. Απλά παίρνουμε τα κονδύλια που υπολείπονται για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη που το χρειάζονται. Όταν το πρόγραμμα λήξει, τελείωσε έληξε. Μετά μπορούμε να δούμε την κατάσταση, να συλλέξουμε πληροφορίες, να δούμε αν έχει νόημα να δοθούν περισσότερα κονδύλια, τι είναι δυνατόν, τι όχι. Δεν πρόκειται για ε, αυτοματισμούς εδώ, δημιουργεί αυτοματισμός, ούτε για ε, παρατάσεις ε, SAE. Αυτό το λέω για λόγους σαφήνειας και γι' αυτό μάλιστα έχουμε υποβάλει τις σχετικές τροπολογίες. Και θεωρώ λοιπόν πως το πρόγραμμα αυτό αξίζει τη στήριξή μας. Με τις τροπολογίες μας εξάλλου προσπαθήσαμε να μην αυξήσουμε τη γραφειοκρατία, αλλά το αντίθετο, με τις τροπολογίες μας προσπαθήσαμε να δώσουμε μία ε, σαφή γραμμή, να ε, δημιουργήσουμε όσο το δυνατόν λιγότερη γραφειοκρατία. Και εδώ έχω και μία παράκληση για τους συναδέλφους. Στις τροπολογίες σας μην ε, επεκταθείτε, μην οδηγηθούμε σε μια έκθεση που θα εμποδίσει ε, τις χώρες να χρησιμοποιήσουν αυτά τα κονδύλια, μην ε, υποβάλλετε τροπολογίες που θα αναφέρουν υπερβολικούς ελέγχους, υποβολές αναφορών κτλ, συγκεκριμένες προϋποθέσεις για το ποια έργα θα στηρίζονται, μην ε, κάνουμε την έκθεση μια έρημο αχανή, γεμάτη προϋποθέσεις και όρους. Μην κάνουμε τα πράγματα δηλαδή δύσκολα για τα κρατημέλη. Ας τα βοηθήσουμε για να χρησιμοποιήσουν ε, τα κονδύλια αυτά και να τα ζητούν όσο το δυνατόν ευκολότερα. Είναι κονδύλια τα οποία ε, τα κράτη θα χρησιμοποιήσουν για ε, μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα διακρίνονται από απόλυτη διαφάνεια. Γι' αυτό λοιπόν θα Χαίρομαι πάρα πολύ αν οι συνάδελφοι ακολουθήσουν τις, ε, τη γραμμή που ακολουθήσαμε εγώ και ο κύριος Φανίστελρο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά είχαν να πούν οι συνεισηγητές. Τώρα θα δώσω το λόγο στους και όδης εισηγητές της Επιτροπής μας. Ε, κυρία Τόμασιτς δεν είναι εδώ νομίζω. Δεν τη βλέπω στην αίθουσα. Ο κύριος Γιάκοφτσιτς λοιπόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για ε, την ε, ηγεσία που δείξατε σε αυτή την υπόθεση και ε, για το γεγονός ότι μας επιτρέψετε να Έχουμε αυτό το πρόγραμμα, συνδέεται και με την πολιτική συνοχή και με την οικονομική πολιτική και επιτρέπει την ε, αυξημένη συνεργασία και αποτελεσματικότητα. Ε, έτσι θα αρχίζει και καλύτερα το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Βεβαίως θα πρέπει να βλέπουμε κάθε φορά τις ιδιαίτερες ανάγκες Ε, των κρατών μελών, ε, τις ιδιαίτερες ενδεχομένω απαιτήσει και τα αιτήματα. Εν πάση περιπτώσει θέλω να ευχαριστήσω τον Λάμπερτ και την Κωνσταντσε ε, για τη συνεισφορά τους μέχρι τώρα και πρέπει να πω ότι είχαμε κάποιες επιφυλάξεις αρχικά ε, ε, ως ε, προς τη νέα αυτή πρόταση. Έχω όμως την αίσθηση ότι το πρόγραμμα στήριξη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων πηγαίνει σωστή κατεύθυνση και μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια καλή συμφωνία. Βεβαίως, θέλω να υποστηρίξω τις τροπολογίες των δύο συνσηγητών γιατί εγγράφονται στη συνέχεια των όσων εμείς πάγια ζητούμε και αυτό που θέλουμε να αναδυθεί από την Επιτροπή μας. Ελπίζω το συντομότερο τώρα να στορθούμε στη δουλειά, να το φέρουμε σε αίσιο για να τελειώνουμε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για όλα τα κράτη-μέλη, αλλά και για τη λειτουργία την ίδια των συστημάτων χρηματοδότησης. Άρα Ελπίζω να μπορέσει να αρχίσει το συντομότερο τριμερής διάλογος για να μπορέσουμε εκεί να υπερασπιστούμε τις θέσεις μας. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω τον κύριο Μαρζέ, ούτε την κυρία Ρέντκε. No, they're not present. Απουσιάζουν ε, η κυρία Νταμάτο. Grazie, Ευχαριστώ. Πρόεδρε, αυτή είναι η δεύτερη ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά το πρόγραμμα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων κατόπιν της συνάντησης με τον Επίτροπο. Ευχαριστούμε τους δύο συνεισηγητές. Έχουμε αυτό το σχέδιο κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οπότε και τώρα ε, μπορούμε να ακούσουμε τις απόψεις των υπολείπων και να τα συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα. Τώρα θα ήθελα να σταθώ σε κάποια σημεία τα οποία βελτιώνουν ε, το νομοθέτημα, την ε, ε, παράγραφο 10 και συγκεκριμένα την ε, τροπολογία 6, από εδώ που φαίνεται το πόσο σημαντικό είναι να ενημερώνει το Κοινοβούλιο, επίση την τροπολογία 10, όπου εκεί ορίζεται η πηγή της χρηματοδότησης για αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο είπαμε ότι δεν θα πρέπει να αποτελέσει προηγούμενο για μελλοντικά νομοθετήματα. Πάντως, για μας το ζουμί είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει, γιατί υπάρχει για το άρθρο 5, το που λέγει 29. Εδώ υπάρχει μια αντίφαση, λέει για κάποιου τομεί. Εκεί λέει ότι θα πρέπει να καλυφθούν οι στόχοι του εργασία και εδώ έχουν προσθέσει οι συνεισηγητέ ότι θα πρέπει να υπάρχει κατάρτιση πολιτική ε, εργασίας, κάποια συστήματα γενικη προνοια συστήματα βοήθεια από πλευρά δημόσια υγεία, μετανάστευση σύνορα και αναφέρουν και τη συνοχή, συναδελφοί. Το πρόβλημα όμως είναι ότι οι διαφορετικές ε, μεταρρυθμίσεις είναι τελείως άσχετες με την συνοχή. Μιλάμε για 143 εκατομμύρια τα οποία θα πρικοδοτήσουν το πρόγραμμα και αυτό μου φαίνεται αστείο γιατί προβλέπεται πέρα για Κύπρο και Ελλάδα έχουμε τον ορισμό του κανονισμού και σχετίζει το πρόγραμμα με την κοινωνική πρόνοια, αγορά εργασίας, της ιδιωτικοποίησης υπηρεσιών ε, και επίσης μιλά για παιδεία και κατάρτιση και εκπαίδευση αλλά σε Ελλάδα, Κύπρο και Πορτογαλία τα προγράμματα μεταρρύθμισης δεν βοηθάνε ούτε την ανάπτυξη ε, ούτε την οικονομία των κρατών μελών. Αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι αυξάνουν τους ε, ανέργους, παροξύνουν τις κοινωνικές ε, ανισότητες και αυτό αφορά εκατομμύρια πολιτών. Να επομένως εδώ η Ελλάδα, η Ελλάδα που γίνει απικία της ε, Τρόικας και εκεί μιλάμε για ανεργία των νέων 30-55%. Έχουν χαθεί τόσες θέσεις εργασίας. Μιλάμε 270% ε, αυτή την ύφεση και ε, επίσης έχει χαθεί κάθε υπηρεσία όσον αφορά τη δημόσια υγεία. Έχουμε την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ που τα έχει συζητήσει αυτά και μιλάει, έχει συζητηθεί η κρίση στα κράτη-μέλη και επίσης μιλούμε για την συρρήγνωση των δαπανών για την οικονομική, δημοσιονομική προσαρμογή σε Ελλάδα και Κύπρο. Και εδώ όμως οδηγούμεθα σε περιθωριοποίηση των μη προνομιούχων που έχουν όμως δικαίωμα σε παιδεία και σε κατάρτιση. Εμείς ως πολιτική ομάδα είμαστε κατά αυτών των διαρθωτικών μέτρων, τα οποία είναι επιζήμια. Θα έπρεπε να έχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα από την πολιτική αυτή, από την πολιτική συνοχή. Επομένως θεωρούμε ότι έχουμε όλα τα μέσα πολιτικής, έχουμε τα επιχειρησιακά, περιφερειακά και εθνικά προγράμματα. Έτσι μπορούμε να βοηθήσουμε τις περιφέρειες και διοικητικά. Το πρόγραμμα 14 με 20 θα υπάρξει αυτό το πρόγραμμα το οποίο θα είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Και θα έχουμε τη μεταρρύθμιση μετά το 2020 που θα βοηθήσει περισσότερο την πολιτική συνοχή. Thank you. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Μαρζέ, ο οποίος ήρθε από άλλη επιτροπή ε, στην οποία ψήφιζαν. Ε, έχετε το λόγο κύριο Μαρζέ. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Το συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά είμαστε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος που είχαμε ψηφοφορίες για την κύρωση της ε, Συμφωνίας των Παρισίων. Για ε, το θέμα αυτό που μας απασχολεί τώρα. Ε, όταν είχε έρθει η Επίτροπος, συζητήσαμε μαζί της για κάποια προβλήματα σχετικά με τη συνοχή. Γιατί είχαμε εκφράσει κάποια έλλειψη κατανόηση για το γεγονός ότι παίρνουν κονδύλια από τα περιφερειακά ταμεία ε, από τη συνοχή για να τα δώσουν στην τεχνική βοήθεια. Χαιρόμαστε που έχει αυτό κάπως αποκατασταθεί, αλλά πρέπει να σας πω και το εξής. Παραμένουν κάποιες δυσκολίες Νομίζω ότι εδώ πρόκειται για κάποια χειραγώγηση της πολιτικής συνοχής που τη μεταχειρίζονται ε, για ε, να ε, εξυπηρετήσουν άλλους στόχους που δεν έχουν πάντα μεγάλη σχέση με τη συνοχή και την περιφερειακή πολιτική. Εδώ προκειμένου σκέφτομαι τους στόχους του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Τούτου λεχθέντων βεβαίως Πιστεύω ότι πρέπει να υποστηρίξουμε τους εισηγητές ε, στην προσπάθειά τους να ενισχύσουν τη τεχνική βοήθεια προς τα κράτη-μέλη για να επιτευχθούν οι στόχοι της περιφερειακής πολιτικής. Θα πρέπει πάντα να φροντίζουμε και να επαγρυπνούμε έτσι ώστε να είναι η τελευταία φορά αυτοί που έρχονται να πάρουν από τη συνοχή κονδύλια για να εξυπηρετήσουν άλλους στόχους. Η Επιτροπή μας σε Περιφερειακής Ανάπτυξης θα πρέπει να τα λέει αυτά και να τα διατρανώνει, όπως το κάναμε και προς τον Επίτροπο όταν είχε έρθει εδώ. Thank you. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε την ανταλλαγή απόψε. Ο κ. Ολμπρίχτ, ο οποίος είναι συντάκτης νομοδότησης της Επιτροπής Προϋπολογισμών για το ίδιο θέμα. Παρακαλώ. Καλά τα λέω. Ε, ε, Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω πως συμμερίζομαι και εγώ την άποψη ότι το θέμα είναι ε, κάτι που δεν είναι καθόλου απλό, παρότι τα κονδύλια δεν είναι πολλά. Η πρώτη εντύπωση που αποκομίζω είναι ότι υπάρχει μια τάση να χρησιμοποιούνται κονδύλια από τη συνοχή για άλλους λόγους. Και εδώ επιστρέφουμε στη συζήτηση για την μακροοικονομική αιρεσιμότητα της πολιτικής συνοχής είναι κάτι που το έχουμε ξανασυζητήσει. Τώρα βλέπουμε τις συνέπειες. Είναι αποτέλεσμα των συστάσεων αναχώρα. Και βέβαια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να δώσει κίνητρο στα κράτη-μέλη να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους ή τουλάχιστον τις κατευθυντήριες γραμμές των συστάσεων αναχώρα. Και ίσως ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να χρησιμοποιηθούν άλλοι πόροι. Το θέμα όμως είναι το πώς θα γίνει και επίσης το ότι αυτό είναι κάτι το προαιρετικό και όχι κάτι το υποχρεωτικό. Το θέμα λοιπόν είναι αν τα κράτη-μέλη θα ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιηθεί αυτό το μέσο για να κάνουν ε, μεταρρυθμίσεις στις χώρες τους. Αν θα ζητήσουν δηλαδή την συνδρομή των εμπειρογνωμόνων της Κομισιόν. Και αυτό είναι και η αδυναμία του ε, προγράμματος ε, αυτού. Από την άλλη, δεν μπορούμε να ξαναγκάσουμε τα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα με κονδύλια από το Ταμείο Συνοχή, να κάνουν μεταρρυθμίσει. Ε, επικροτώ βέβαια τι προσπάθειε των συνεισηγητών εάν τα κονδύλια αυτά πράγματι πηγαίνουν από την τεχνική υποστήριξη των ταμείων στην οχή συστάσει συστάσεις αναχώρα. Αυτό, ε, όπως ε, το είπαν και άλλοι, είναι επικίνδυνο. Είναι μια χειραγώγηση της κατάστασης. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη διασύνδεση στην με την πολιτική συνοχής. Διότι η πολιτική συνοχή επηρεάζει πραγματικά πολλούς διαφορετικούς τομείς και πολιτικές. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει τα κονδύλια αυτά να μείνουν εντός της πολιτικής συνοχής για να δείξουμε ότι ε, ότι χρησιμοποιούνται για τις συστάσεις αναχώρα. Καλώς μέχρι εδώ, όμως δεν πρέπει να τα πηγαίνουμε αλλού, γιατί μετά το 2020 θα αλλάξουν τα πράγματα και δεν πρέπει να δημιουργηθεί προηγούμενο για το μέλλον. Διότι στην περίπτωση αυτή τα κονδύλια του Ταμείου Συνοχής θα είναι ένα αποθεματικό για να τα χρησιμοποιούν οι άλλοι κατά το δοκούν. Επιτροπή μας συμφώνησε με το να χρησιμοποιηθούν αυτά τα κονδύλια από την πολιτική συνοχή, αλλά ας δούμε που πηγαίνουν. Από την Γενική Διεύθυνση Ρέγγιο σε άλλη ε, σε άλλο θεσμικό όργανο. Γι' αυτό λοιπόν τι σχέση έχει αυτό με τις συστάσεις αναχώρα. Θα έπρεπε λοιπόν να ε, πούμε ναι υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν ε, ισχυροί δεσμοί με την πολιτική συνοχής για να γίνει αυτό. Στην Επιτροπή Προϋπολογισμών θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το ίδιο, να στηρίξουμε δηλαδή αυτή τη γραμμή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Νοβάκοφ έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όταν προτάθηκε αυτό το πρόγραμμα, πολύ πριν παρουσιαστεί στο Κοινοβούλιο, άρχισα να το παρακολουθώ και να παρακολουθώ και τις εξελίξεις. Και παρέμειναν κάποια αναπάντητα ερωτήματα, έχω να πω. Γι' αυτό λοιπόν μην θεωρήσετε με αυτά που θα πω ότι είμαι ξεκάθαρα υπέρ ή κατά της πρότασης, αλλά προσπαθώ να είμαι αντικειμενικός πρέπει να δούμε αποτελέσματα, τα αποτελέσματα που θα ε, έρθουν. Με τον προϋπολογισμό αυτό, τα κράτη-μέλη έχουν περίπου στη διάθεσή τους 5 εκατομμύρια ευρώ το καθένα. Πιστεύετε εσείς πραγματικά ότι θα κάνουν τη διαφορά αυτά τα 5 εκατομμύρια ευρώ θέλω να δω τι θα γίνει με 5 εκατομμύρια ευρώ στη Γαλλία ή στη Γερμανία, αν θα καταφέρει να γίνει κάτι, να αλλάξει κάτι. Πρέπει να συμφωνήσουμε ότι εάν χρησιμοποιούμε χρήματα από το Ταμείο Συνοχής για άλλο, ε, ότι δεν θα στρώσουμε το δρόμο έτσι για να γίνει αυτό ε, και την επόμενη χρονιά και την μεθεπόμενη χρονιά και να γίνει συνήθεια. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 4 ετών. Νομίζω πως όλοι καταλαβαίνουμε εδώ στην αίθουσα ότι για να έχουν αποτέλεσμα κάποια προγράμματα συνοχής θέλουν πολλά περισσότερα χρόνια. Αυτό φαίνεται και από την αγορά, φαίνεται και από, τον, το εκπαιδευτικό σύστημα, φαίνεται πόσο διαρκούν οι μεταρρυθμίσεις και σίγουρα δεν είναι μόνο τέσσερα χρόνια. Συμφωνώ από την άλλη ότι χρειάζονται μεταρρυθμίσεις ε, σε ορισμένα κράτη-μέλη. Όμως υπάρχουν ήδη ε, προγράμματα επιχειρησιακά για τεχνική υποστήριξη που ε, γίνονται αυτή τη στιγμή, βρίσκονται να εξελίξει. Εάν επιτρέψουμε λοιπόν να γίνει αυτή η επικάλυψη, τότε θα θολώσει το τοπίο, θα αυξηθεί η γραφειοκρατία. Δεν θα ξέρουμε πού είναι τα ωριά μας που αρχίζουν τα χωράφια των άλλων. Και το πρόβλημα είναι ότι παρέχεται λοιπόν αυτή η δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης στα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη όμως θα τη γιατί εγώ πραγματικά θέλω να δω τι θα γίνει. Δεν είμαι αρνητικός, ωστόσο πιστεύω πως η πρόταση αυτή χρειάζεται πολύ περισσότερες διευκρινήσεις. Διαφορετικά αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά από αυτό που διαβάζω. Υπάρχουν άλλα από πίσω. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα πολύ περισσότερες λεπτομέρειες, επεξηγήσεις, για να καταλάβουμε το γενικότερο πλαίσιο του προβλήματος. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Νίλσεν έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχω ήδη λάβει μέρο στη ζήτηση. Μιλώ αγγλικά γιατί δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη μητρική μου γλώσσα, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει διερμηνία από τη γλώσσα μου. Οπότε, ο συνήθως ο κύριος Φανίστηλ Ρόε και η κυρία Κρέλ επιτελούν έργο αξιόλογο και εστιάζουν την προσοχή εκεί που πρέπει και από τη χώρα μου τι έχω μάθει. Ότι, ότι πάντοτε κάθε απόφαση, κάθε ό,τι σχετίζεται με το Περιφερειακό Ταμείο δημιουργεί μεταξύ των εκεί αρχών ε, μεγάλο καυγάδι ότι θα γίνουν τα κονδύλια για την τεχνική βοήθεια. Οι τοπικές αρχές των ίδιων πολιτών λένε ότι χρειάζεται να υπάρξουν αυτά τα κονδύλια για να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους συνεταιρισμούς, τους διάφορους φορείς για να μπορέσουν να καλυφθούν από το πρόγραμμα. Χρειάζονται τα στιγμή τη βοήθεια και λέει η κυβέρνηση όμω όχι, πρέπει να χρησιμοποιηθεί η πρικοδότηση για τα, τα έργα και τις πολιτικές της κυβέρνησης και κερδίζουν τη μάχη και έτσι γίνεται κάθε μία πενταετία. Οπότε θεωρώ ότι και αυτή τη φορά πρόκειται να δοθεί μάχη και ο Υπουργό Οικονομικών θα αγωνιστεί για να μπορέσει να πάρει αυτό την πρικοδότηση τεχνική βοήθεια. για πει ότι ναι υπάρχει αυτό το πρόγραμμα ακόμα και αν δεν χρειάζεται αλλά χρειαζόμαστε τα χρήματα και δεν θα μπορέσουν να κερδίσουν τον αγώνα οι τοπικέ αρχέ Να, πώ είναι τα πράγματα στη Σουηδία. Η πρόεδρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Κρέλ, έχετε το λόγο. Ακριβώς αυτό εννοούσα. Ότι στην αρχή θα πρέπει να κοιτάξουμε και μόνοι μας και χρειάστηκε να δούμε και μόνοι μας ε, τι θα έπρεπε να κάνει το νέο αυτό μέσο. Και οι δύο τελευταίοι ομιλητές ε, το κατέδειξαν σαφώς. Υπάρχουν ακόμα τέτοιες παρεξηγήσεις. Το συγκεκριμένο εργαλείο, το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν έχει σκοπό να ενισχύσει, ξέρω εγώ, τη μεταρρύθμιση των τραπεζών κάπου, στην Τσεχία ας πω, ξέρω εγώ, να χρηματοδοτήσει και να διεξαγάγει. Δεν είναι γι' αυτό το λόγο φτιαγμένο. Αλλά εάν η τσεχική δημοκρατία θέλει, σε περίπτωση που θέλει να κάνει μια μεταρρύθμιση, λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωραία. Αν θέλετε τεχνική βοήθεια, αν θέλετε τεχνική υποστήριξη, θα σας στείλουμε έναν ε, αρμόδιο εμπειρογνώμονα για τα τραπεζικά, δεν ξέρω από πού, από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ή από κάπου αλλού, που μπορεί να σας βοηθήσει πώς θα το οργανώσετε. Η μεταρρύθμιση ίδια είναι υπόθεση του κράτους και βεβαίως χρειάζεται περισσότερο από μια τετραετία. Αλλά δεν είναι ε, ο στόχος ούτε το νόημα του νέου αυτού μέσου, του νέου εργαλείου να χρηματοδοτεί τη μεταρρύθμιση. Τεχνική βοήθεια παρέχει και εξασφαλίζει. Και γι' αυτό από την αρχή δεν έχουν μοιραστεί τα 142 εκατομμύρια τόσα θα πάρει Σουηδία, τόσα θα πάρει Βουλγαρία, τόσα θα πάρει Γερμανία. Όχι. Είναι ε, μόνο μετά από αίτημα. Εγώ υποθέτω ότι η Σουηδία δεν πρόκειται ποτέ να καταφύγει σε αυτό, γιατί πιστεύω ότι λειτουργεί πολύ καλά ως χώρα. Ε, ούτε η Γερμανία θα το ζητήσει. Αλλά θα μπορούσα να φανταστώ ότι ξέρω εγώ, η Κροατία θα χρειαστεί να καταφύγει σε αυτό ή η Βουλγαρία για να ζητήσει τεχνική βοήθεια και δημιουργείται έτσι ο σύνδεσμος. Λέμε, εντάξει, η τραπεζική μεταρρύθμιση δεν έχει μεγάλη σχέση με την πολιτική συνοχή. Ας είναι εξαίρεση. Αλλά αν κάνουμε μια μεταρρύθμιση στα εργασιακά ή αν κάνουμε μια μεταρρύθμιση στο σύστημα υγείας, αυτές είναι αρμοδιότητες που ε, συγχρηματοδοτούνται από την πολιτική συνοχή. Και υπάρχει και πληθώρα παραδειγμάτων και πληθώρα αναγκών όπου μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει και να καταφύγει σε αυτή την βοήθεια. Γιάννης, έχεις απολύτως δίκιο για τον καυγά, για την τεχνική βοήθεια στα κράτη-μέλη. Παντού ο ίδιος είναι. Απλώς τίθεται το εξή ερώτημα. Δεν αφαιρούμε τίποτα από καμία χώρα μέλος. Απλώς τα χρήματα που είχαν προβλεφθεί για τεχνική βοήθεια. Παίρνουμε 142 εκατομμύρια και θα πρέπει να είναι σαφές ότι υπάρχει μεγάλη σχέση με την πολιτική συνοχή ε, και δημιουργείται και μια κατάσταση έκτακτη δεν θα αποτελέσει προηγούμενο και ποτέ δεν μπορεί κανείς να αναγκαστεί να κάνει κάτι. Είναι πραγματικά σε θελούσια βάση και επίση θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι εάν ένα κράτο μέλος δεν το αξιοποιεί, δεν το χρησιμοποιεί, δεν σημαίνει ότι θα του ωφεληθούν ή θα του κουπούν τα κονδύλια συνοχή. Δεν υπάρχει τέτοια αυτόματη σύνδεση. Ελπίζω να έρθουν τροπολογίες που να ενισχύσουν αυτά που λέμε, αλλά προς αυτή την κατεύθυνση θέλουμε να στραφούμε από κοινού. Thank you. It was like an answer. Ευχαριστώ. Μάλλον απάντηση σε ερωτήσεις συναδέλφων. Το λόγο έχει η κυρία Ρέντκε. Thanks a lot. And sorry. Ευχαριστώ. Συγχωρείτε που άρχισα, αλλά και εσείς νομίζω αρχίσατε να το κοβεντιάσετε πιο νωρίς από ό,τι έπρεπε, οπότε δεν μπόρεσα να είμαι εδώ για mm. όλη τη συζήτηση. <laughs> Sometimes uh, we have uh, Uh, especially if coming from smaller groups, you have. Uh, για τις μικρότερες ε, πολιτικές ομάδες υπάρχει πρόβλημα. Τέλος πάντων, ε, χαίρομαι πολύ που κάνουμε τη συζήτηση. Για να σας πω περίπου πώς θέλουμε να διαμορφωθεί η κατάσταση από πλευράς της δικής μας ομάδας. Τώρα αυτή η συζήτηση έχει ευρύτερη σημασία ε, γιατί εδώ εμπλέκονται περισσότερε πολιτικέ ομάδε, όσο και αν εμεί έχουμε το ρόλο του συντονιστή, η Επιτροπή Περιβάλλοντο, αλλά θα πρέπει να αλλάξουμε την πρόταση της Επιτροπής. Θα πρέπει επίσης να πολιτικοποιήσουμε το θέμα, να μην μιλάμε μόνο για τι ε, τεχνικές λεπτομέρειες, γιατί θα μπορούσε αυτή η υπόθεση να είναι ένα μέσο σημαντικό και τα κράτη-μέλη να μπορούν να βοηθηθούν στη διαχείριση και να αξιοποιούν περισσότερο τις πολιτικές συνοχής και να είναι πιο δυναμική η προσέγγιση και να πιάνουν τόπο οι ευρωπαϊκές επενδύσεις. Όπως είναι όμως σήμερα η πρόταση της Επιτροπής, επειδή έχει κινδύνους. Γιατί αν δεν αξιοποιηθεί αυτό το μέσο ε, τις ε, μεταρρυθμίσεις ε, και θέλει να κατευθύνει τα κρατημέλη σε συγκεκριμένη κατεύθυνση για τις επενδύσεις, τότε ελοχεύει ο κίνδυνος κατάχρησης αυτού του μέσου πολιτικής, αυτού του εργαλείου. Οπότε εμείς αυτό που θέλουμε είναι να επιμείνουμε, να επιμείνουμε για την πολιτική συνοχή γιατί είδαμε τι έγινε σε Ελλάδα και Κύπρο. Δεν τα πήγαν και τόσο καλά τέτοιε προτάσεις όσον αφορά την αξιοποίηση των ε, διαρθωτικών ταμείων. Δεν τα πήγαν πολύ καλά σε όλα τα μέτωπα. Άρα θα πρέπει να ε, ασχολούμαι και με άλλα θέματα και όχι μόνο με την οικονομική διακυβέρνηση. Κάτι άλλο σημαντικό για μας Θέλουμε μία διαδικασία πιο σφαιρική για τις προτεραιότητες των επενδύσεων για να πιάσουν περισσότερο τόπο αυτή η πόρη για να μπορέσει να εμπλακεί κοινωνία των πολιτών, τοπικές αρχές βέβαια και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Άρα θα πρέπει ρητός να αναφερθεί ότι οι πόροι θα διατεθούν και για αυτούς τους εμπλεγωμένους. Επίσης, θέλουμε να δούμε πώς θα καλυφθούν οι δυνατότητες της διοίκησης, οι περιφερειακοί εμπλεκόμενοι και κάποιοι ντόπιοι εμπειρογνώμες. Μην δοθεί η εντύπωση ότι αυτό είναι καπέλωμα από πάνω από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τα κάτι μέλη. Πάντως, θεωρούμε πολύ θετικό το ότι συνεργαστήκαμε με τους συζητητές και τους σκιώδες συζητητές. Νομίζω ότι αυτό το κείμενο αξίζει πιο βαθύ προβληματισμό και να συνεργαστούμε με τις άλλες πολιτικές ομάδες ούτως ώστε όλα αυτά που σας είπαμε μπορέσουμε να τα περάσουμε. Η Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε. Θέλει άλλο το λόγο. Όχι. Κύριος Φανίστελ θέλει τώρα να απαντήσει κάποιες από τις ερωτήσεις. Ναι, να επαναλάβω ότι καταρχάς η διαδικασία είναι ανοιχτή. Έχουμε τις συνδεδεμένες επιτροπές, έχουμε τη δυνατότητα να υποβάλουμε τροπολογίες και θα προσπαθήσουμε να ε, δώσουμε τη δυνατότητα στα κράτη-μέρη που έχουν ανάγκη να καταφέρουν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους. Η Επιτροπή μας είναι η αρμόδια Επιτροπή. Αυτό είναι σαφέστατο. Και σε πολλές τροπολογίες φαίνεται η ανάγκη που υπάρχει για πληροφορίες που ζητάμε ε, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, η διαδικασία να είναι διάφανη κτλ. Ο Επίτροπος θα έρχεται στην Επιτροπή μας να μας ενημερώνει. Είναι ε, λοιπόν η διαδικασία ανοιχτή, σταθερή, διάφανη και ε, ένα μέτρο προαιρετικό. Δεν υποχρεώνεται κανείς να ζητήσει σύνδρομη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν υποχρεώνουμε κανέναν να πάρει κονδύλι από ένα ταμείο και να τα πάει στο άλλο. Αυτό φαίνεται στο έγγραφο, φαίνεται στο σχέδιο έκθεσης και για παράδειγμα η τροπολογία 15 μιλάει για συνέργειες. Και όπως είπε και η κυρία Κρέλ, το ζητούμενο είναι ε, να ε, κάνουμε τα πράγματα με καλύτερο τρόπο χωρίς ε, προβλήματα. Το είπατε και εσείς και οι συνάδελφοι άλλωστε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι πολύ σημαντικές και οι τροπολογίες που υποβάλλεται. Ο στόχος όμως ποιος είναι. Ο στόχος είναι πολιτικές να μένουν στον στόχο τους, να μην παρεκτρέπονται. Υπάρχουν συγκεκριμένα κονδύλια τα οποία πρέπει να διτίθεται για συγκεκριμένους σκοπούς. Όμως, πρέπει να φροντίσουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έρχεται, να μας ενημερώνει και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες εκεί που μπορεί. Δεν θα ανοίξουμε με αυτήν την πρόταση το κουτί της Πανδώρας, δεν θα χάσουμε για πάντα τα κονδύλια από την συνοχή. Είναι ένα κείμενο το οποίο μπορούμε να υπερψηφίσουμε ή να καταψηφίσουμε, να το τροποποιήσουμε. Το είπε και η κυρία Κρέλλα άλλωστε. ο στόχος μας είναι η ανάκαμψη των ε, κρατών μελών που το έχουν ανάγκη και ακούστηκε ότι αυτή η πολιτική σκοτώνει, δολοφονεί, διαλύει τις θέσεις εργασίας, δεν δημιουργεί καινούργιες. Το είπε η κυρία Νταμάτο. Και πρέπει να φροντίσουμε λοιπόν να ακουστούν όλες οι γνώμες ε, και πρέπει να φροντίσουμε αυτή η εικόνα που μας έδωσε η κυρία Ανταμάτο να μην γίνει πραγματικότητα. Τώρα, ε, κύριε Ομαρζέ, κάνατε πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα και ρωτήσατε και τον Επίτροπο κιόλα ε, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Τον πιέσατε και αναγνώρισα την πολιτική συνοχή ως ένα από τα σημαντικότερα μέσα που έχουμε για την στήριξη και τα ταμεία επίσης που συνδέονται με την συνοχή. Αλλά ας δούμε αν θα δημιουργηθούν συνέργειες εδώ, ας δούμε τι αποτελέσματα θα έχουν και μετά ας περάσουμε στο επόμενο βήμα. Εσείς φυσικά ευχαρίστω να υποβάλλετε τις τροπολογίες σας γιατί στόχος μας είναι να μας στηρίξετε εν τέλει. Ευχαριστώ. Εάν δεν θέλει κάποιος άλλος το λόγο, θα ήθελα εγώ να πω μερικά λόγια για το θέμα. Καταρχάς να ευχαριστήσω τους συνεισηγητές, την κυρία Κρέλ και τον κύριο Βανίστελ Ρόι για τη δουλειά που έχουν κάνει και τη στάση που τήρησαν, έτσι ώστε να δημιουργηθούν αυτές οι συνέργειες ανάμεσα σε αυτό που προτείνει η Επιτροπή και στις αρμοδιότητες της ε, δικής μας Επιτροπής. Διότι είναι πολύ δύσκολο να ε, αναλάβουμε εμεί ω Επιτροπή Περιφερειακή Ανάπτυξης την ευθύνη για αυτό το θέμα και είναι καθήκον μα επομένως να προτείνουμε μια λύση η οποία θα είναι ε, ισορροπημένη και θα συνδέει την οικονομική διακυβέρνηση, την ανάπτυξη και τις ε, θέσεις απασχόλησης με το ρόλο της πολιτικής συνοχής. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για την προσέγγιση που υιοθετήσατε και ελπίζω να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας. Διότι άκουσα από τους εισηγητές το εξής, ότι στην αρχή υπήρχαν πολλά ερωτήματα, υπήρχαν αμφιβολίες, τώρα μειώθηκαν αυτές οι αμφιβολίες, διότι οι εισηγητές μας κατάφεραν να βρουν μια λύση. Ελπίζω λοιπόν οι συζητήσει να οδηγήσουν σε αποτελέσματα, διότι πρόκειται για τη δημιουργία ενός νέου μέσου που δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει. Καθήκον μας όμως είναι να προσπαθήσουμε να λειτουργήσει όσο το δυνατόν καλύτερα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να το συζητήσουμε, να κάνουμε τροποποιήσεις, να σκεφτούμε πώ αυτό το μέσο θα είναι πιο αποτελεσματικό και ε, θα ε, συνδέεται περισσότερο με την πολιτική συνοχή. Εγώ από την πλευρά μου θα κάνω ό,τι μπορώ για να δημιουργηθεί ένα καλό κλίμα στις συζητήσεις. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Ρίεν, εκπρόσωπο της Επιτροπής των Περιφερειών, η συγγήτρια για το θέμα αυτό. Έχετε το λόγο. Κυρία Όλγα Σρίεν, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο και ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους που ε, θα με ακούσουν ε, να πω δύο λόγια ως εισηγήτρια της Επιτροπής των Περιφερειών. Τον Απρίλιο εγκρίναμε τη γνωμοδότησή μας. Ήδη ε, είχαμε προτείνει 20 συγκεκριμένες νομοθετικές τροπολογίες στην Επιτροπή Περιφερειών όλοι θεωρούμε αυτή την ευκαιρία πραγματικά πολύτιμη έτσι ώστε να υπάρξει συνεργασία μεταξύ της δικής σας Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών για ένα μέτρο που όπως είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε είναι πάρα πολύ καινούριο και θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε μια μεγάλη πρόκληση για την ευρωπαϊκή οικονομική ολοκλήρωση. Θα δούμε πόσο αποτελεσματική είναι και πόσο δημοκρατική η Ένωση οι δημόσιες αρχές και μεταξύ αυτών η ΟΤΑ θα ε, δείξουν πόσο μπορούν να παίξουν ε, ρόλο στις αυτοτικές μεταρρυθμίσεις. Κάναμε μια συζήτηση σήμερα που αυτό το αποδεικνύει περίτρανα. Η Επιτροπή των Περιφερειών ε, δέχεται και εγκρίνει καταρχήν το πρόγραμμα αυτό υποστήριξης τεχνικής βοήθειας πάντα σε θεντοντική βάση και κατόπιν αιτήματος του κάθε κράτους μέλους. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Παρ' όλα αυτά, το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής νομίζω χρειάζεται κάποιες διευκρινήσεις και θα πρέπει να φροντίσουμε να έρθουν οι διευκρινήσεις αυτές. Η βελτίωση της διοικητικής και θεσμικής ικανότητα κάθε κράτος μέλους αφορά και την κεντρική κυβέρνηση αλλά και τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης. Και αυτό θα πρέπει να είναι στον πυρήνα του προγράμματος για τα κράτη που το επιθυμούν. Θυμίζω ότι 40% ε, των συστάσεων αναχώρα για το 2016 αναφέρονται σε αυτές τις δυνατότητες της δημόσιας διοίκησης ε, που είναι ή δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει περιφερειακές προκλήσεις και αυτό αφορά και την τοπική αυτοδιοίκηση. Παρ' όλα αυτά, η υποστήριξη αυτή θα πρέπει να έχει να κάνει με τομεί δράση όπου είναι συντρέχουσε οι αρμοδιότητε ε, των κρατών μελών και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν το έχει ξεκαθαρίσει αρκετά στο κείμενό τη αυτό το συγκεκριμένο. Άρα το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι προσβάσιμο για τη ΣΟΤΑ βάσει ε, τη ε, κατανομή των εξουσιών σε κάθε χώρα ε, και τις αρμοδιότητες. Άκουσα ότι υπάρχουν δυσκολίες στη Σουηδία και το καταλαβαίνω, αλλά θα πρέπει και οι συστάσεις αναχώρα που συχνά απευθύνονται στις ΟΤΑ ε, θα πρέπει να ε, βρίσκουν κάποια αντανάκλαση και ανταπόκριση. Αυτά όλα και χαιρόμαστε γι' αυτό εκφράζονται ξεκάθαρα στη δική σας έκθεση. Η Επιτροπή Περιφερειών θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα στρατηγικό έγγραφο ενιαίο για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη βελτίωση της θεσμικής και διοικητικής ικανότητας της δημόσιας διοίκησης σε κάθε επίπεδο διακυβέρνησης. Έκανε και το ελεκτικό συνέδριο κάποιες παρατηρήσεις για την τεχνική βοήθεια στην Ελλάδα, καθώς επίσης και το σχέδιο έκθεσή σας, ένα ενιαίο λοιπόν στρατηγικό έγγραφο που θα πρέπει να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα του προγράμματος διότι θα επιτρέψει καλύτερο και πιο αποτελεσματικό συντονισμό με τα προγράμματα τεχνικής βοήθειας που υπάρχουν ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, στα δικαιούχα κράτη. Επίσης θα πρέπει να έχουμε μεγάλη ε, δέσμευση των κονδυλίων και συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών εκτός από την τοπική αυτοδιοίκηση και των κοινωνικών εταίρων. Αυτό είναι εκ των όνων Κάνευ για την ε, επιτυχία του προγράμματος. Και είναι επίσης τελείως απαραίτητο έτσι ώστε να αυξηθεί η εμπιστοσύνη, να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ κρατών μελών που το επιθυμούν, ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ε, των άλλων κρατών. Επίση, το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να είναι πιλωτικό και να αξιολογηθεί εν ευθέτω χρόνο για να δούμε αν θα ε, χρειαστεί να παγιωθεί και να μονιμοποιηθεί. Και απαντάει αυτό σε κάποια ερώτησή Σε περίπτωση που θεωρηθεί κάτι τέτοιο σκόπιμο, μπορεί να χρειαστεί ένα ταμείο ε, ε, που να χρηματοδοτείται από ιδίου πόρου. Θα πρέπει να δούμε αν αυτό είναι επιθυμητό, εφικτό ή απαραίτητο. Είναι γεγονό ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί ε, η κατάσταση αυτή που επικρατεί σήμερα μόνο προσωρινή και μεταβατική μπορεί να είναι. Και κατά τα άλλα είμαστε αντίθετοι με τον να ανοίξει τρόπο και ένας δρόμος υποταγής ε, της πολιτικής συνοχής ε, στι συστάσεις αναχώρα. Τι θα γίνει δηλαδή, θα εξχεδιάζεται η πολιτική συνοχή σαν ένα εξάμεινο είναι ξεχωριστή πολιτική, αναγνωρισμένη και κατοχυρωμένη από τις συνθήκες και χαίρομαι που ε, λέτε κι εσείς εδώ αυτά που είπαμε στην Επιτροπή Περιφερειών. Ελπίζουμε η συνοχή τελικά να μην πέσει θύμα σε αυτή την υπόθεση. Σας ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή σας και που με ακούσατε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank you. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, η Πρόεδρος. Έχουμε της Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην κυρία Μέρη Μακάρθια, αλλά και την κυρία Αν Κέρστινγκ Μίλε. Ποια θέλει πρώτη το λόγο, για να μιλήσετε και οι δύο. Hello, um, I'm Mary McCarthy from... Εδώ εργάζομαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είμαι διευθύντρια στην υπηρεσία για τις ε, διευθυντικές μεταρρυθμίσεις και σας ευχαριστούμε για την έκθεση. Και περιμένουμε διακάζω να προχωρήσει η συζήτηση και είμαστε διαθέσιμοι για οποιαδήποτε διευκρίνηση θα θέλατε για οποιοδήποτε σημείο που θεωρείτε δεν είναι σαφές. Ευχαρίστως να σας τα εξηγήσουμε. Στη διάθεσή σας. Yes, if I may. Uh, I'm from the Regional Policy. Ε, εργάζομαι στην Γενική Διεύθυνση της Περιφερειακής Πολιτικής και επιβεβαιώνω αυτά τα οποία είπε η συνάδελφος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνεργαζόμαστε στενά και εμεί επίσης στη διάθεσή σας για ό,τι διευκρίνηση και ενημέρωση επιθυμείτε. Ευχαριστούμε. Εμεί ευχαριστούμε λέει ο Πρόεδρος. Ε, βέβαια και περιμένουμε να συνεργαστείτε, χρειαζόμαστε τη συνεργασία μαζί σας όσον αφορά τη διαμόρφωση τη τελική εκδοχή του κειμένου και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να το έχουμε συντάξει σύντομα. Ευχαριστούμε και καλή τύχη για την υπόλοιπη διαδρομή. Τώρα, η προθεσμία των τροπολογιών. Σας προτείνω να είναι το μεσημέρι της Τετάρτης 14 Ενάτου. Συμφωνείτε? Δεκάτη Τετάρτη του μήνας. Τετάρτη. Αυτή είναι η καταληκτική ημερομηνία για και εδώ κληρώθηκε η συζήτηση όσον αφορά το θέμα αυτό. Συνεχίζουμε. Έχουμε την έκθεση της κυρίας Μπρέσον που αφορά την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. One of the Είναι ένα από τα αγαπημένα μας θέματα στην Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής. η Οικονομική Επιτροπή αλλά και η Επιτροπή των Προπολογισμών έχουν συντάξει μια έκθεση όσον αφορά το πρώτο έτο τη δραστηριότητα αυτού του Ταμείου για τι Στρατηγικέ Επενδύσει. Και η κυρία Μπρέσο είναι η ε, συντάκτρια τη γνωμοδότηση για τη δική μα Επιτροπή και έχει ετοιμάσει την έκθεση για τη δική μα Επιτροπή που αφορά αυτό το πρώτο έτο λειτουργία. και σα προτείνω καταληκτική ημερομηνία για τι τροπολογίε τη έκθεση και πάλι το μεσημέρι της 14ης Σεπτεμβρίου. Οπότε και για αυτόν τρόπο να μπορέσουμε να ψηφίσουμε τον Οκτώβριο στην συνεδρίαση. Κύριε Μπρέσο, έχετε το λόγο για να μπορείτε να μας εισηγηθείτε το σχέδιο κειμένου. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και στα Ιταλικά ευχαριστώ και όπως γνωρίζετε εν τη αυτή περιπτώση πρόκειται για κάποια γνωμές. Συμπάθατε με λίγο μισό αυτό. Σας παρακαλώ λέει πρόεδρος κυρίες και κύριοι. Κυρίες και κύριοι, όποιος θέλει να αποχωρήσει να το πράξει ησύχως. Και πάλι ευχαριστώ πρώτα λέει η κυρία Μπρέσο. Σας έλεγα ότι όπως θα γνωρίζετε έχουμε σε αυτή την ε, περίπτωση τη συναρμοδιότητα, ή μάλλον την κυρίω αρμοδιότητα τη Επιτροπή Προπολισμού και τη Οικονομική Επιτροπή. Αλλά έχουμε και εμεί αυτή την έκθεση που αφορά την λειτουργία αυτή τη πρώτη φάση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Οπότε είναι η δική μα συμβολή πολύ σημαντική, διότι ε, παρά το ότι επανειλημμένα είπαμε ότι θα πρέπει να συμβάλλουμε στην οικονομική και περιφερειακή συνοχή και θα μπορούμε να έχουμε περισσότερη προσθετικότητα και περισσότερες συνέργειες ε, μεταξύ των ε, διαρκικών ταμείων. Το θέμα είναι ότι τη σήμερα ημέρα επί τη βάση των στοιχείων που έχουμε, που έχουμε λέγω, δίνουν ένα θετικό μήνυμα όσον αφορά την εξέλιξη αυτού του, αυτούς της πολιτικής. Ε, υπάρχουν κάποια project, έχουν χρηματοδοθεί αρκετά, επομένως τα πράγματα κινούνται. Πάντως, ε, σαφώς προκύπτει ότι από την άλλη μεριά ε, έχουμε θέμα με τις συνέργειες μεταξύ των διαδοτικών ταμείων και του ΕΤΣΕ, του ΕΦΣΕ, σύμφωνα με το πλάνο Γιούνκερ. Ακόμα, επομένως, ε, δεν πάνε καλά αυτές οι συνέργειες. Οπότε εμείς πρώτα πρώτα το τονίσαμε αυτό. Δεν υπάρχουν συνέργειες παρά τις προσπάθειες που γίνεται. Οπότε και εμείς εδώ καλούμε την ΕΤΕ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις εθνικέ, Κεντρικές ε, Τράπεζες, ε, τις τράπεζες αναπτυξιακές τέλο πάντων, να στηρίξουν τους επενδυτές και έτσι να επιταχυνθεί ο ρυθμός αυτών των συνεργειών. Βέβαια, είναι πάρα πολύ χρήσιμο για αυτά τα έργα και προγράμματα να υπάρχει η δυνατότητα, να υπάρχει αρκετή κρατική χρηματοδότηση που να συνοδεύει τις τραπεζικές ε, χρηματοδοτήσεις, κάτι το οποίο ισχύει για το Ταμείο Στατικών Επενδύσεων. Και έτσι αυτό είναι, κάνει και καλύτερο κλίμα για την πολιτική συνοχή. Πρώτα πρώτα θέλω να σου πω ότι θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Πρέπει να υπάρχουν εγγυήσει τέτοια συνεργασία όσον αφορά τα εμπλεκόμενα ε, τραπεζικά ιδρύματα για του εμπλεκόμενα φορεί όπω η ΕΤΕ κλπ. Είναι θέμα στρατηγική. Δεύτερον, κάτι το οποίο συνδέεται με αυτό το οποίο μας απασχολεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εδώ πέρα το, το πάνω χέρι, θα πρέπει να δούμε και τον γεωγραφικό χαρακτήρα αυτών των ε, έργων και προγραμμάτων. Διότι προς το παρόν το πρόγραμμα Juncker επικεντρώνεται σε κάποιες χώρες που ίσως δεν χρειάζονται αυτή την προσθετικότητα τόσο ώστε να μπορέσουν να έχουν τις επενδύσεις. Η προσθετικότητα τελικά είναι κάτι πολύ σημαντικό αλλά όχι τόσο για κάποιε χώρε που ήδη έχουν δυνατότητε επένδυση. Άρα, αυτό το οποίο θέλουμε εμεί είναι να ληφθεί υπόψη μια γεωγραφική ισορροπία, να υπάρχει μια τέτοια συνέργεια των διευθυντικών ταμείων. Και κυρίω αυτό αφορά τις ε, χώρε ή τι περιφέρειες με λιγότερη ανάπτυξη. Οπότε, έχουμε και κάποιου έργα και προγράμματα διασυνοριακά και αυτά θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να συνδέονται με τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές, αυτά τα οποία έχουμε τονίσει στην πρώτη εκδοχή του κειμένου μας, ότι μέχρι τώρα δεν έχουμε αποτελέσματα σε αυτό το μέτωπο. Άρα να ληφθεί υπόψη αυτού του είδους η γεωγραφική ισορροπία στο πρόγραμμα Juncker Επίσης το ότι θα πρέπει να υπάρχει συνέργεια με τις πολιτικές συνοχής Επίση να λαμβάνεται υπόψη ο ισενεργειακό χαρακτήρα, ο υπερεθνικό, να θέλετε, αυτών των έργων. Πολύ σημαντικό. Και αυτό θα πρέπει οι αρμόδιε επιτροπέ να το λάβουν υπόψη. Αυτό το οποίο λέμε και επίση οι Τράπεζα επενδύσουν Άλλο σημείο τώρα. Εκεί όπου επισημαίνουμε στην έκθεση ότι θα πρέπει να προσέξουμε να δούμε τι γίνεται από πλευρά θεματική με αυτά τα έργα. Κάτι το οποίο θα πρέπει να συνάδει με τους στόχους της αναπτυξιακής πολιτικής. Πρόκειται για κάποιους στόχους που είναι παλιοί και είναι κάποιες επενδύσεις χρήσιμες που δημιουργούν περιβάλλον δημιουργίας, ανάπτυξης και απασχόλησης. Άλλο τώρα, το τονίζουμε, είναι το ότι θα πρέπει να ε, επιλεγούν κάποια μέτρα χρηματοδότησης με αξιοπιστία και διαφάνεια. Έτσι θα πρέπει να γίνεται η επιλογή των έργων. Δεν έχουμε τώρα διαφάνεια, θα πρέπει να την αποκτήσουμε. Α, επίσης, και για την επιλογή αυτών των έργων χρειάζονται σχέσεις όχι μόνο με τις κρατικές, αλλά με τοπικές και περιφερειακές αρχές Πρόκειται για έργα που αφορούν ε, τη, τα περιφερειακά και το έτσε. Άρα θα πρέπει να ενισχύσουμε τις ε, περιφερειακές και εθνικές πλατφόρμες. Και έτσι να καταλήξουμε σε συνέργειες. Οπότε να έχουμε ε, τέτοια έργα που όπως είπαμε να καλύπτονται από τα εν λόγω ταμεία διαθωτικά ταμεία, πλάνο Juncker, ε, αυτά τα έργα θα πρέπει να εξαιρούνται από τους υπολογισμούς του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και για τα κράτη και χωριστά για περιφερειακές και τοπικές αρχές. Επίσης, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εμπλακεί. Είναι σημαντικό θα πρέπει να αναβαθμίσουμε την αρμοδιότητά μας παρακολούθησης και εποπτείας ε, όλες αυτές τις υποθέσεις. Το πλάνο Γιούγκερ θα εξελιχθεί, ενδεχομένως θα τροποποιηθεί, αλλά ε, βέβαια αυτό θα πρέπει να συνδευτεί από χρηματοδοτική υποστήριξη. Δεν θέλουμε να υπάρξουν επενδύσεις που θα αποκλίνουν. Να έχουμε κάποια στρατηγική σε αυτές τις επενδύσεις εν ώψη του Ευρώπη 2020. Ούτε αυτό υπάρχει προς το παρόν. Αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό να συμβεί. Να έχουν συνοχή, συνέπεια, λογική αυτές οι επενδύσεις. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα να δώσουμε το λόγο στους σκιώδεις Πόλτσακ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μπρέσο για την παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης που πιστεύω ότι καλύπτει όλες τις ε, σημαντικές ε, λειτουργίες για την ομαλή ε, εξέλιξη του σχεδίου Juncker. Ταυτόχρονα όμως η έκθεση δεν αποφεύγει τα αμφιλεγόμενα και επίμαχα ζητήματα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μπρέσο για την ειλικρίνεια και την αυθύτητά της. Τα μία αυτά έχουν κινητοποιήσει πόρους ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέτος το καλοκαίρι με μία δήλωσή της δήλωσε ότι η έλλειψη κινητοποίησης οφείλεται σε, ε, στα κράτη-μέλη. Και ο, το κύριο εμπόδιο είναι το διοικητικό άχθος και υπερβολική γραφειοκρατία. Ε, πιστεύω πως αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γι' αυτό θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Μπρέσο αν έχει ίδια κάποιες προτάσεις και ιδέες γι' αυτό, έτσι ώστε να τη συμπεριλάβει στην έκθεσή της. Επίσης προσωπικά θεωρώ πως είναι ε, εξαιρετικά σημαντικό να ε, δούμε τι ακριβώς έργα στηρίζει το ΕΦΣΥ. Και πιστεύω πως δεν είναι απόλυτα σαφές ε, αν αυτά τα έργα έχουν υψηλό κίνδυνο ή όχι. Και πιστεύω πως τα έργα τα οποία στηρίζουμε είναι έργα υψηλού κινδύνου. Είναι λοιπόν ένα σημαντικό θέμα το οποίο πρέπει να ασχοληθεί αυτή η Επιτροπή, διότι η ιδιαιτερότητα των, ε, του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων είναι ότι ακριβώς στηρίζει έργα τα οποία είναι υψηλού κινδύνου. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να αναρωτηθούμε εάν αυτή η προϋπόθεση ερεσιμότητας ε, τηρείται. βλέπω ότι υπάρχει έλλειψη στήριξης στα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, αλλά νομίζω πως αυτό δεν ήταν κάτι εσκεμμένο από την εισηγήτρια. Ίσως όμως η έκθεση να μπορούσε να ε, τονίσει περισσότερο την σημασία αυτών των ταμείων στρατηγικών επενδύσεων. Τα ταμεία αυτά ε, ίσως ε, θεωρηθούν ανταγωνιστικά και πως θα θυσιαστούν επενδύσεις για να εγγυηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση την επιτυχία του ΕΦΣΥ. Θα έπρεπε λοιπόν να ενδιαφέρει όλους εμάς που είμαστε μέλη της Επιτροπής η διατήρηση αυτών των ταμείων και γι' αυτό πρέπει να στέλνουμε ένα ισχυρό μήνυμα και στα άλλα θεσμικά όργανα θεωρώ πως η σημερινή ανταλλαγή απόψεων είναι μία πρόγευση του τι θα ακολουθήσει. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μπρέσο για τη δουλειά που έχει κάνει. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μάσιτς δεν νομίζω πως έχει έρθει. Επόμενος και ο εισηγητής εκ μέρους της ε, ομάδας Άλτερ είναι υποφανόμενη. Θα ήθελα λοιπόν και εγώ να πω δύο λόγια για την έκθεση της κυρίας Μπρέσο. Ευχαριστώ πολύ κυρία. Λοιπόν, κύριε Μπρέσο για τη γνωμοδότησή σας. Και θα ήθελα να τονίσω ότι έχουμε καλά αποτελέσματα. Είδαμε ότι το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων έχει δώσει θετικά αποτελέσματα δεδομένων των δημοσιονομικών περιορισμών στα κράτη-μέλη. Έπρεπε λοιπόν να πλουστευτούν οι διαδικασίες και να ζητήσουμε ε, να είναι συμπληρωματικά, να έχουν συμπληρωματικό ρόλο τα ταμεία, ε, τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία. Αυτό όμως θεωρώ πως θα κινητοποιήσει τον χρηματοπιστωτικό και τον ιδιωτικό τομέα και θα μεγαλώσει τις θετικές επιπτώσεις, θα οδηγήσει σε αύξηση ε, και ανάκαμψη της οικονομίας. Είναι λοιπόν στόχος μας να στηρίξουμε έργα που θα φέρουν προς τη θέμενη αξία και θα ενισχύσουν και τον Ευρωπαϊκό, την Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Πλατφόρμα Επενδύσεων. η συνδρομή της ε, ΕΤΕ νομίζω πως δεν καταφέρνει να φτάσει σε περιφερειακό επίπεδο, να στηρίξει έργα σε περιφερειακό επίπεδο και το συμβουλευτικό έργο θα έπρεπε να φτάνει μέχρι τους τελικούς δικαιούχους. Και τα έργα εκείνα που καταφέρνουν να δημιουργήσουν συνέργειες ανάμεσα στα δύο αυτά ταμεία. Γι' αυτό και θα στηρίξω την γνωμοδότηση της εισηγήτριας. Επίσης, θέλουμε να δούμε και μία επιγραμμική πλατφόρμα η οποία θα συνδέσει τους επενδυτές με τα επενδυτικά έργα. Αυτή λοιπόν η διαδικτυακή πύλη πιστεύω πως θα έπρεπε να είναι περισσότερο ορατή για να επιτρέψει την προσέλκυση κεφαλαίου που είναι πολύ σημαντικό για το Ταμείο στρατηγικών Επενδύσεων άλλωστε. Τώρα, πώ μπορούμε να συνδυάσουμε το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων με τα διαθερωτικά και επενδυτικά ταμεία, έτσι ώστε να γίνουν πραγματικά μεγάλε επενδύσει. Εδώ απαιτούνται τα κατάλληλα μέσα για να πλουστεύσουν αυτήν την ε, σύνδεση. Και αναφέρομαι ιδιαίτερα στη συνεργασία ανάμεσα στα διάφορα μέσα, το συντονισμό και τις συνέργειες ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και στα Διευθυντικά και Επενδυτικά Ταμεία. Τέλος, να τονίσω πόσο σημαντικό είναι να βελτιώσουμε την ε, πρόσβαση του κοινού στην πληροφορία, να μαθαίνουν οι πολίτες τις επιτυχίες του Ταμείου, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει αναπαρκής ενημέρωση, ακόμα και για εμάς, εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο, παρότι ε, η αρμοδιότητά μας είναι να παρακολουθούμε την επιτυχία της ε, εφαρμογής των του Ταμείου στα έργα. Πρέπει λοιπόν να μπορούμε να αξιολογήσουμε τα έργα αν είναι υψηλού κινδύνου, αν χρησιμοποιούν τα κονδύλια με το σωστό τρόπο, εάν αυξάνεται η ορατότητά τους στο κοινό και αν υπάρχουν αυτές οι συνέργειες ανάμεσα στα δύο ταμεία. Αυτά λοιπόν ήθελα να πω με το ρόλο της καιόδου εισηγήτριας και τώρα θα δώσω το λόγο στην Μαρτίνα Μίχελ η οποία λείπει και θα, θα δώσω λοιπόν το λόγο στην κυρία Ράινκε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη γνωμοδότησή της. Όλοι συμφωνούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα για την Επιτροπή μας πώς μπορούν να συνδυαστούν τα κονδύλια αυτά με το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ε, χαιρόμαστε πάρα πολύ που το συζητούμε αυτό το θέμα και ταυτόχρονα ε, ακούστηκε και μια ανησυχία, εκφράστηκε μια αγωνία με την οποία συμφωνώ. Ε, τι γίνεται με τη συνέπεια και τη συνέχεια των επενδύσεων αυτών. Τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Πολλές είναι οι προκλήσεις που πρέπει να ξεπεράσουμε και τα προβλήματα Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε μια κριτική ματιά και προσέγγιση στη σημερινή εφαρμογή ε, και απορρόφηση των κονδυλίων, όχι επειδή δεν χρησιμοποιούνται αυτά τα κονδύλια, αλλά θέλουμε να βελτιωθεί η ε, χρήση τους και να πιάσουν τόπο. Γι' αυτό παραμένουμε πάρα πολύ επιφυλακτικοί και διστακτικοί σε σχέση με την παρούσα κατάσταση. Τι άλλο που θα θέλαμε να ενισχυθεί στην πρόταση είναι το εξής. Η αρχή της προσθετικότητας είναι κάτι που θέλουμε να έχουμε ισχυρότερη θέση από πλευράς της Επιτροπής μας. Και ένα δεύτερο, που ρωτάμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι γίνεται για την προστασία για τις πρώτες απώλειες. Ε, στην αρχή μας είπανε ότι το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων θα τα κάλυπτε αυτά ε, τις πιο ε, επισφαλής ε, δόσεις των επενδύσεων. Τώρα φαίνεται ότι αλλάζει αυτό και επομίζεται το βάρος κάποιο διαρθρωτικό ταμείο. Ανησυχούμε πολύ και θα πρέπει η Επιτροπή μας να το πει αυτό, να μην υπάρξει αυτή η αλλαγή και η ανατροπή. Και κάτι άλλο που έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο, πιστεύω, στη δημόσια συζήτηση για το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων γενικά, είναι η περίφημη μόχλευση. Πώς μπορούμε δηλαδή να αυξήσουμε τα κονδύλια αυτά και τη μόχλευση σε σχέση με τα όσα βλέπουμε σήμερα, γιατί υπολείπεται φυσικά το ποσό των προσδοκιών και των εξαγγελιών. Γι' αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε στη γνωμοδότησή μας. Και κάτι που έχει τεράστια σημασία εδώ είναι η διαφάνεια στα προγράμματα αυτά και πώς μπορούμε να τα διαφημίσουμε περισσότερο, να γίνουν πιο γνωστά και να οικοδομηθεί και εμπιστοσύνη και να έρθουν και ιδιωτικέ επενδύσεις προσβλέπω σε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με ανταλλαγή απόψεων και έντονη και διαφωνίες και συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Η κυρία Νταμάτο. Ναι, έχουμε υπόψη μας το ότι προσπαθεί να βελτιώσει τα πράγματα η έκθεση όμως θα πρέπει να δούμε το ότι δεν εξυπηρετεί αυτό το πρόγραμμα. Θα έχουμε τα νέα έργα της ΕΤΕ που θα πρέπει να υποστηρίζουν. Αλλά όμως με τι κριτήρια, πώς γίνεται η επιλογή. Είπαμε ε, ότι έχει προτεραιότητες η Επιτροπή, αλλά χρειάζεται να δούμε πώς προκύπτουν αυτές οι προτεραιότητες με συγκεκριμένο τρόπο, πώς γίνονται οι αξιολογήσεις, πώς γίνεται η επιλογή. Έχουμε εδώ διάφορα στοιχεία ε, για να ε, ε, αξιοποιηθεί το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα των επενδύσεων. Όμως δεν έχουμε στα χέρια μας συγκεκριμένα το πώς θα πιάσει τόπο το εύση. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις εγγύσεις, τι θα γίνει με τα ορυκτά κάψιμα. Θα έχουμε βιοαέριο, βιομάζα, αλλά δεν λέγεται τίποτα όσον αφορά την ε, αυτονομία και την αυτάρκεια με τις τράπεζες πώς θα υποστηρίξουν τις ΜΜΕ να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε περισσότερη κερδοσκοπία και φούσκες. Κάτι άλλο τώρα από το έτσι το ότι πολλαπλασιάζονται τα έργα για τα οποία τα στοιχεία δεν αποκαλύπτονται, ενώ εγκρίνονται τα έργα. Πρόκειται εδώ για τον δημόσιο κορβανά. Έτσι θα στηριχθεί το ΕΦΣΕ. Ε, άρα θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια για κάθε δράση του ταμείου αυτού. Να μπορεί ο κόσμος να ξέρει πού πάνε τα λεφτά του. Τι μπορεί να κάνει το κοινοβούλιο να υποπτεύσει, να ελέγξει πώς θα ασκήσουμε αυτήν την αρμοδιότητα εάν δεν έχουμε πληροφορίες. Έρχεται και μας λέει δύο-τρία λόγια τη μία μέρα, δύο-τρία την άλλη κάποιος επίτροπος. Θέλουμε όμως συγκεκριμένα στοιχεία. Ακριβώς αυτά που ζητούμε. Θα πρέπει ο, κόσμος να ξέρει ότι έχουμε ανάπτυξη, προστασία του περιβάλλοντος, να ενισχυθούν οι ΜΜΕ, να πάνε για καινοτομία. Και το πλάνο Γιούνκερ θεωρούμε ότι δεν είναι η απάντηση στις πραγματικές υπάρχουσες ανάγκες. Σας ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Και συνεχίζουμε. Ο κύριος Τσέλερ, παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Λοιπόν, αν κάποιος θέλει να μάθει ποια είναι τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στα πλαίσια αυτού του Ταμείου ε, Στρατηγικών Επενδύσεων, μπορεί να το μάθει στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Εκεί αναγράφονται όλα τα έργα, όλα τα projects και είναι μεγάλη η ποικιλία των έργων και των προθέσεων που ε, χρηματοδοτεί. Πολλά αεολικά πάρκα offshore, στο Παρίσι μεγάλες εταιρείες ε, κατασκευής ε, ε, διαμερισμάτων που θέλουν εξηγιά διαμερίσματα κατοικίες. Είναι προγράμματα γεωργικά, όλα εγκάρσια. Δεν έχουν πάρα πολύ μεγάλη σχέση όλα αυτά με την πολιτική συνοχή όμως. Και αν δω τις προτάσεις της κυρίας Μπρέσο και δεν κάνω λάθος στην ερμηνεία, θα ήθελα μια ε, πολύ πιο ισχυρή μορφή συντονισμού ε, του σχεδίου Juncker, του Ταμείου Juncker στρατηγικών επενδύσεων με την ε, Τράπεζα Επενδύσεων. Θέλω να προειδοποιήσω, είναι τελείω διαφορετικέ φιλοσοφίε η διαρθρωτική πολιτική και αυτό που αποσκοπεί το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Δηλαδή, το ΕΦΣΙ τι θέλει, καλύπτει τους κινδύνους με δημόσια χρήματα που έχουμε βγάλει από τον προπολογισμό για να προσελκύσει και να κινητοποιήσει ιδιωτικέ επενδύσεις που κατά τα άλλα δεν πηγαίνουν οι ιδιωτικέ επενδύσει ε, στην έρευνα και την καινοτομία, στη γεωργία και αλλού, επειδή έχει κίνδυνο και δεν του καλύπτουν το κίνδυνο και δεν πάνε οι ιδιώτε να τα επενδύσουν. Οπότε αυτό είναι ο στόχο του όλου εγχειρήματο. Τώρα, ποιο πρόβλημα έχουμε. Έχουμε χρήματα από το Δημόσιο Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα, αλλά και από αλλού, από την διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη. Τα πήραν από εκεί αυτά τα λεφτά, αλλά τα υπόλοιπα τα διεκπερώνει μια τράπεζα με βάση τραπεζικά κριτήρια. Εμείς θα πρέπει να δώσουμε μια μάχη έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν τελειώσει ε, και λήξει ο πρώτος γύρος του ΕΦΣΥ να μας φέρουν μια δήλωση, μια αναφορά, τι έγινε με τα λεφτά που προέρχονται από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό και πώς τα έχουν διαχειριστεί οι τράπεζες. Είναι κατεξοχήν τραπεζική λοιπόν η διεκπαιρέωση. Και τώρα ε, έχουμε και την ερώτηση. Το 2017 ε, υπήρχε περιορισμός, δηλαδή ναι, μέχρι το 2017 το ΕΦΣΙ θα παραταθεί ε, αυτή η διάρκεια. Αν γίνει αυτό χρειαζόμαστε νέο χρήμα φρέσκο για να χρηματοδοτήσουμε και νέα έργα σύμφωνα με τη φιλοσοφία του παρόντος ταμείου. Δεν έχει λυθεί από πού θα βρεθούν. Εγώ δεν πιστεύω ότι οι συνάδελφοι από τις μεταφορές ή από την έρευνα και την επιστήμη θα είναι ακόμα διατεθειμένοι από το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα να δώσουν και άλλα κονδύλια για τα προγράμματα του ΕΦΣΥ. Ή ότι θα ξαναπάμε στο Connecting Europe να πάρουμε λεφτά. Ούτε πρέπει, ούτε πρέπει να το θέλουμε κάτι τέτοιο. Αλλά για να υπάρχει μια συνοχή ανάμεσα στην πολιτική συνοχή και τη διαρθρωτική και το ΕΦΣΥ, θα ήταν σκόπιμο να πούμε ότι υπάρχουν κάποια κονδύλια από τα διαστατικά προγράμματα που μπορούμε να τα χρηματοδοτήσουμε, να τα δώσουμε για τη χρηματοδότηση με το ΕΦΣΥ. Όμως εκεί είναι ολιστηρό το έδαφος και δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουμε και πώς θα έχει η πολιτική συνοχή μετά το 2020 και η διαρθρωτική πολιτική. Και δεν ξέρουμε και πού θα καταλήξουμε μήπως πέσουμε και σπάσουμε τα μούτρα μας. Θα πρέπει να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν και η Τράπεζα Επενδύσεων τι έχει γίνει μέχρι τώρα στα πλαίσια του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων να ζητήσουμε και απόδειξη τι γίνεται με τα χρήματα που έχουμε διαθέσει εμείς από τον περιπολογισμό έχουν πιάσει τόπο έχουν προσελκύσει μάλλον ιδιωτικές επενδύσεις αξιόλογες. Μέχρι τώρα διαβάζω ότι εντάξει προγραμματίζεται να έρθουν και άλλες ιδιωτικές επενδύσεις, τάζουν δηλαδή ότι θα έρθουν κάποια λεφτά πέρα από εκείνα που έχουμε βάλει εμείς και η Τράπεζα Επενδύσεων. Να το κρατήσουμε αυτό λοιπόν και να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια, πώς θα εξελιχθεί η πολιτική συνοχή και η διαρθρωτική που έχει άλλη ιδεολογία, άλλη φιλοσοφία με κοινοτικά κονδύλια από τον κοινοτικό γνωσιακό προπολογισμό σε συνεργασία με τις αρχές τοπικής ή περιφερειακής αυτοδιοίκησης ή και με τις εθνικές αρχές που είναι επίση δημόσιο για να ενισχυθεί η ανάπτυξη, η οικονομία και βεβαίως και η κοινωνική συνοχή να ε, προωθηθεί. Αυτό είναι κάτι τελείω διαφορετικό από τη φιλοσοφία και τις προθέσει του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Και θα πρέπει να τα έχουμε ξεχωριστά μέχρι να ξεκαθαρίσει πού το πάει αυτό το ταμείο και τι συνέχεια θα δοθεί. Τουλάχιστον αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βαλκάρθερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ να συγχαρώ την εισηγήτρια για το εξαίρετο έργο της στην γνωμοδότηση αυτή η κυρία Μπερέσο πάρα πολύ εύστοχα έθιξε όλα τα προβλήματα για την εφαρμογή του Ταμείου Στατηγικών Επενδύσεων για την συμπληρωματικότητα, προσθετικότητα, συνέργειες όσον αφορά τις στρατηγικές αυτές επενδύσεις τα τα ταμεία και τα ταμεία επενδύσεων. Εγώ θέλω να σταθώ σε αυτή την προσθετικότητα. Θα πρέπει το ταμείο να χρησιμοποιηθεί για κάποια έργα που δεν θα χρηματοδοτηθούν από τα ταμεία επενδύσεων και τα διαρθρωτικά. Δεν θα υποκατασταθούν αυτά τα ταμεία. Απλώς έτσι θα έχουμε περισσότερες επενδύσεις. Επίσης είναι σημαντικό αυτό το ταμείο τελικά να μην χρηματοδοτήσει κάποια έργα που θα χρηματοδοτηθούν από τον ιδιωτικό τομέα. Να χρηματοδοτηθούν μόνο τα έργα τα οποία δεν έχουν χρηματοδότηση και χρειάζονται αυτή την έξτρα χρηματοδότηση. Γι' αυτό και χρειάζεται να υπάρξει γεωγραφική ισορροπία, όπως είπε η συγκήτρια και να προωθήσουμε διασυνοριακά έργα που δίνουν προς θεμήνη αξία. Ε, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, λέει Πρόεδρος. Κύριε Μπουστινάρο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα αρχίσω με ευχαριστίες. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Mercedes Πρέσο για την καταπληκτική της ε, εργασία, το σχέδιο αυτογνωμοδότησης. Πώς να το πω, είναι πραγματικά μια πάρα πολύ εύστοχη εικόνα σε αυτό που μας είχαν παρουσιάσει πάρα πολύ ρόδινο ορισμένοι επίτροποι και τώρα το, και θυμάστε το ευρωπαϊκό αφήγημα στην αρχή ότι θα ήταν ένα μέγα εργαλείο αν όχι ή πανάκια για να λύσει όλα μας τα προβλήματα και τι λέει η πραγματικότητα, καμία σχέση με αυτό το αφήγημα και με ε, όσα μας έταζαν οι προσδοκίες. Πρώτον, ε, είναι γεγονό και το επιβεβαίωσε και η Μερσέντε και όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό που λείπει είναι η στρατηγική φύση των επενδύσεων. Μέσω αυτού του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων όλες. Γιατί επενδύουμε σε τραμ ή σε μόνωση κτηρίων με στρατηγικές επενδύσεις. Τι είναι αυτό, στρατηγική επένδυση, το τραμ και η μόνωση των κτηρίων καλύπτει ε, καμιά ρηψοκίνδυνη επένδυση, όχι. Είναι για να απορροφηθούν τα κονδύλια ή να τα πάρουμε επειδή είναι φτηνά λεφτά. Δεν μας αρκεί αυτό. Δεύτερον, αν κοιτάξουμε τη γεωγραφική κατανομή των επενδύσεων, τι διαπιστώνουμε. Ορισμένοι από εμά θα θυμόμαστε πάρα πολύ καλά τη μάχη που δώσαμε ε, στη διευκόλυνση νέοντας στην Ευρώπη. Διότι μας είχαν πει από την αρχή ότι όποιος προλάβει Όποιος έρθει πρώτος θα πάρει ε, το Ταμείο Στρατηγικών επιδίσεων. Είμαστε μεν παρόντες. Δεν θα αναφερθώ στη Ρουμανία, θα αναφερθώ στην Πολωνία. Η Πολωνία είναι πρωταθλήτρια στον τρόπο με τον οποίο και με πάρα πολύ ευφύ τρόπο μάλιστα απορροφούν τα κονδύλια. Και παρόλα αυτά η Πολωνία σήμερα παίρνει μόνο 80 εκατομμύρια ευρώ. Δεν θα μιλήσω για άλλα μέλη ε, κράτη-μέλη της συνοχής. Και έχω μια πάρα πολύ πικρή ερώτηση. Sorry κιόλα, αλλά τα κράτη-μέλη της συνοχής συνεισφέρουν, βάζουν 10 δισεκατομμύρια ευρώ στο Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Και όταν έρχεστε και μας λέτε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν έχουμε γεωγραφικά κριτήρια, δεν έχουμε γεωγραφική ισορροπία και κατανομή, τότε εγώ έχω μεγάλο πρόβλημα. Διότι τα χρήματα πληρώνονται από τις χώρες συνοχής σε χώρες που δεν είναι της συνοχής και παρόλα αυτά φαίνεται ότι είναι πρωταθλητές ε, αντλησής κονδυλίων από το ΕΦΣΥ. Άλλο ζήτημα. Οι συνέργειες πολιτική συνοχής και επενδύσεις από το Ταμείο Στατηγικών Επενδύσεων. υπήρχε ένας όρος επιτακτικός που δεχτήκαμε να πάνε τα λεφτά της συνοχής εκεί, ήταν να υπάρχει συνέργεια με τις επενδύσεις. Να έχουν κάποια συνάφεια με τη συνοχή και τις διαρθρωτικές πολιτικές. Αν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, για ποιο λόγο να δεχτεί τη μεταφορά πιστώσεων αυτή ε, το Κοινοβούλιο και να συνεχίζεται. Γιατί όλοι αναφέρονται στη δυνατότητα όχι μόνο συνέχιση, ε, του ΕΦΣΥ, αλλά και αύξηση μάλιστα της πρικοδότησης. Και ενδεχομένως κάποιοι να εποφθαλμιούν και πάλι το προπολογισμό της συνοχής. Ποιες βεβαιότητες έχουμε, πού είναι οι συνέργειες. Θα πρέπει να είναι ε, με τρόπο μετρήσιμο δεδομένες και όχι με μια ωραία παρουσίαση ότι ότι εντάξει άμα κάνω τραμ θα μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας και η ρήπανση και έτσι είμαι πιο ανταγωνιστικός και λιγότερο ρηπαίνων. Πολύ ωραία αυτά που μας λένε, αλλά καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αυτά εμείς δεν τα χάβουμε, εν πάση περιπτώσει. Και μια πάρα πολύ σοβαρή ερώτηση που έχω. Το, ε, ε, ε, το, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων είναι ένα εγχείρημα, μια άσκηση για να δούμε τι θα υπογίνει με την πολιτική συνοχή. Γιατί από ό,τι φαίνεται οι ίδιοι επίτροποι που έρχονται και μα τα πουλάνε όλα αυτά εδώ τα ρόδινα, είναι εκείνοι που προωθούν την ιδέα ότι το μέλλον της πολιτικής συνοχής θα είναι αυτό. Πάρα πολύ σχετικό με το λεγόμενο σχέδιο Juncker ή ο τρόπος με τον οποίο θα βρεθούν τα κονδύλια για τη χρηματοδότηση της συνοχής και πώς θα πηγαίνουν από τον προϋπολογισμό συνοχής προς τα κράτη-μέλη θα είναι αντίστοιχα. Και κάνουμε έτσι μια άσκηση σε φυσικό μέγεθος ε, για να δούμε πώς θα αναπτυχθεί η πολιτική στο μέλλον. Και πάλι sorry, αλλά εγώ δεν τα χάβω αυτά τα πράγματα. Δεν θα πρέπει τώρα να κάνουν ένα πείραμα για να δούνε πώς θα συνεχιστεί η πολιτική συνοχή και να είναι αυτό. Αν θέλουμε να τη διαφυλάξουμε ως θεμελιώδη παράγοντα, όχι μόνο για την αντιμετώπιση ανισοτήτων, αλλά και γενικότερα για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών, τότε και σε χώρες που είναι καθαροί συνεισφορείς, αλλά και σε χώρες που είναι καθαροί δικαιούχοι, τελειώνω πρόεδρε, ξέρετε μια μελέτη που έκανε η κυρία Βιενκόφσκα, πρώην Υπουργός Εξωτερικών και νυν Επίτροπος, που δείχνει ότι ένα ευρώ από τους καθαρούς συνεισφορείς επιστρέφει από κάθε ευρώ 0,66, τα δύο τρίτα δηλαδή, επιστρέφουν στους καθαρούς συνεισφορείς. Μέσω τεχνογνωσία, συμβουλών, ε, τεχνολογικής υποδομής, εξοπλισμού και από αυτά τα 66, το 76% πηγαίνουν στη Γερμανία ή το 70% που κανονικά είναι η ατμομηχανή, η κινητήρια δύναμη στην Ευρώπη και η μεγαλύτερη βιομηχανική δύναμη. Λοιπόν, α τα δούμε αυτά σοβαρά και να πούμε στην Κομισιόν μην τολμήσετε να παίζετε με το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Και μην νομίζουν ότι ε, θα μας τα κοκουλώσουν και εμείς θα τα χάψουμε έτσι ως κοινοβούλιο. Δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσουμε έτσι ούτε να διερευνούμε για το τι θα γίνει και να πολυδοσκοπούμε το μέλλον της συνοχής να γίνει τράπεζα ή ταμείο επενδύσεων. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Thank you very much, Madam Chair. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ε, να αρχίσω καταρχάς με το ότι η πανάκια που είπατε είναι ελληνική λέξη, κύριε Ποστινάρου. Πιστεύω λοιπόν ότι το Ευρωπαϊκό Τραμείο Στρατηγικών Επενδύσεων δεν είναι πανάκια. Είναι ένα καινοτόμο μέσο που ε, λειτουργεί έτσι, επιφέροντας καινοτομία. Δεν θα συνηθίσω όμως τώρα το πώς λειτουργεί το ΕΦΣΥ, αλλά το σχέδιο γνωμοδότησης εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Θα πάω λοιπόν κατευθείαν στο θέμα. Σύμφωνα με με τις τελευταίες εξελίξεις, όπως μας ενημερώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα επίπεδα απορρόφησης του ΕΦΣΗ είναι κα... στα 110 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα κράτη-μέλη όπως, όπως η Ελλάδα από αυτό το ποσό λαμβάνουν μόνο 535 εκατομμύρια και ε, περιμένουν 1,3 δις να απορροφηθεί. Όπως καταλαβαίνετε το ποσό είναι πάρα πολύ ε, χαμηλό και κάτι δεν πάει καλά. Για μένα υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης για το πώς λειτουργεί το ΕΦΣΥ, έλλειψη πληροφοριών για το πώς δηλαδή μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Θα ήθελα λοιπόν να υποβάλω μια σχετική τροπολογία που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αυξήσει τις προσπάθειες έτσι ώστε να συμπεριληφθούν όλα τα κράτη-μέλη, διότι η Κύπρος ε, είναι, εξαιρείται από αυτήν την ε, διαδικασία και να ενισχυθούν ιδιαίτερα μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διότι εκείνες πρέπει να στηριχθούν. Εκείνες ε, λαμβάνουν μόνο 75 εκατομμύρια και στη δική, μας, στη δική μου χώρα την Ελλάδα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα κονδύλια. Χρειάζεται επίσης ε, να υπάρχει μια αναφορά για το πόσο ο τραπεζικός τομέας συνεργάζεται πολύ στενά με το ΕΦΣΥ διότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτό που έχει ήδη ε, εγκριθεί, όμως να μπορούμε να ε, ενώσουμε τις προσπάθειές μας για να χρησιμοποιήσουμε ό,τι υπολείπεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βανίστηλ Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είμαι ε, λίγο επηρεασμένος και εντυπωσιασμένος από αυτά που ακούω. No way το ένα το άλλο. Πολύ απόλυτα μας τα λέτε. Ε, γνωμοδότηση είναι αυτό για μια έκθεση εφαρμογής ε, για τον προϋπολογισμό. Από αυτά τα No Way θα έρθει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με πρόταση και ε, τούτη την εβδομάδα και την άλλη για παράταση του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Ε, ε εδώ ταράζεστε ας πούμε και φωνασκείτε, αλλά τι θα γίνει. Εδώ ε, μιλάμε για την εφαρμογή ενός ταμείου και τι έκανε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν ξέρω αν μας ακούει, έχει φύγει από εμά και έχει, είναι αλλού τώρα, βρίσκεται πιο μακριά. Όχι μόνο στη Ρέτζη. Αυτά που λέτε εδώ στη Ρέτζη να τα πείτε στις πολιτικές ομάδες. Το αποκλείεται και δεν τα χάβω και no way να τα πείτε στην πολιτική σας ομάδα. Ναι, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει δρόμος, όχι no way, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς διαφορετικά θα το προτείνουμε. Παράδειγμα, ε, οι δημόσιες συμβάσεις. Μπορεί ο καθένας να ε, βάζει λεφτά όπου θέλει, εντάξει είναι τραπεζική διαχείριση. Εμείς είμαστε δεμένοι χειροπόδερα με τις διαδικασίες. Εγώ ε, πραγματικά έχω χάσει το λογαριασμό γιατί μετρούσα πόσα άρθρα δημοσιεύονταν στον τύπο για αυτό το ταμείο. Γύρω στα 50 σταμάτησα γιατί δεν πήγαινε άλλο να μετράω. Και κάθε φορά ε, που κάνει κάτι η Τράπεζα Επενδύσεων φωνάζουμε πω, πω κοιτάξτε σώσαμε την Ευρώπη. Ε, υπάρχει υπερβολή ε, και έχουμε πατήσει και γκάζι, έχουμε επιταχύνει, δεν ξέρω αν υπάρχει 7η, δέκατη ταχύτητα, αλλά κάπως έχουμε αποκοπεί από την πραγματικότητα και από την πραγματικότητα της συζήτησης που κάνουμε εδώ. Δεν καταλήγουμε πουθενά ή καταλήγουμε πάρα πολύ αργά, κατόπιν εορτής. Εγώ ρώτησα πότε θα φέρετε την αξιολόγηση, να ξέρουμε πραγματικά τι γίνεται. Α, είχε προβλεφτεί λέει για το 2017. Πολύ ωραία, θαυμάσια. Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Ωραία, κάνουμε εκθέσεις, εκθεσούλες πρωτοβουλίες, γράφουμε τροπολογιούλες κτλ. Ε, και από εκεί τι θα κάνουμε τώρα. Έχουμε μια λογική παραμία να δω αν μεταφράζεται. Που λέει ότι τα σκυλιά βγίζουν, το καραβάνι περνάει ε, και συνεχίζει το δρόμο του. Ε, και τι γίνεται στις δημόσιες συμβάσεις, τίποτα ούτε μας ακούνε, τίποτα, καμία επικοινωνία, μηδέν. Και οι ηγέτες των πολιτικών ομάδων τι κάνουν, συμφωνούν και τα δέχονται. Ωραία πράγματα. Εγώ θα κάνω την τροπολογία που περιμένετε να κάνω, αλλά σε πολιτικό επίπεδο, στις πολιτικές ομάδες θα πρέπει να συζητηθεί αυτό. Νομίζω ότι εμείς ε, κάπου έχουμε αποτελματωθεί εδώ και άλλοι συνεχίζουν και μας ξεπερνάνε ε, και έχουν προχωρήσει πολύ παρακάτω. Τι πρέπει να κάνουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση αυτή. Θα δώσω τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μετά στην κυρία Βρέσο. Από την Κομισιόν έχουμε την κυρία Φόρετιν Χόπμαγερ από τη Γενική Διεύθυνση ΕΚΦΙΝ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ, σα ευχαριστούμε για την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση, αλλά επίση και για την ευκαιρία που δίνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τοποθετηθεί. Φλόρεντιν Χόπμα, ονομάζομαι, για την ΕΚΦΙΝ και εδώ είναι η από την ε, Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτική. Θα πρέπει να σα πω τα εξή, τόσο ώστε να καλυφθείτε για αυτά που ζητείτε ω ε, βελτιώσει και να σα πω και τι πρόκειται να κάνουμε σε σχέση με την ανακοίνωση της πρώτης έκτου της Επιτροπής πρώτα πρώτα θα ήθελα να σας πω κάποια στοιχεία που αφορούν το έτσι σε αυτό το χρόνο έχουμε κινητοποιήσει 115,7 δις σε κάποιες ε, επενδύσεις 26 κρατομελών και 200.000 ΜΜΕ έχουν ε, ωφεληθεί επίσης, έχουμε καταφέρει να ελκύσουμε και άλλες επενδύσεις, που είναι βέβαια στόχος βασικός. Περίπου 85% των προσδοκομένων επενδύσεων προέρχονται από επενδυτές ε, κρατικούς και από ιδιώτες. Και αυτό το οποίο θέλει το έτσι είναι να μπορέσει να βοηθήσει στην συνοχή τώρα όσον αφορά την γεωγραφική ε, αλλά και την ε, ανατομέα ποικιλία, πολυμορφία, θέλουμε να εξασφαλίσουμε το πώς θα έχουμε περισσότερα έργα από τις χώρες συνοχής. Και έχουμε κάποια εργαλεία προς τούτο, όπως ήδη προαναφέρθηκε πάνω από μια φορά, έχουμε το συνδυασμό της χρήσης του έτσε με άλλες κοινωτικές χρηματοδοτήσεις ιδίω από τα επενδυτικά και διορθωτικά ταμεία. Επίσης η δημοσιοποίηση των καθημερινών γραμμών το Φεβρουάριο του 2016 ήταν απλώς το πρώτο βήμα. Αυτό που τώρα χρειάζεται είναι από τη θεωρία να περάσουμε στην πράξη και έχουμε τώρα την ανακοίνωση της πρώτης ε, έκτου και εκεί. Ρητά προβλέπεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕΤΕ πρόκειται να έχουν κάποια έργα τα οποία θα είναι συγκεκριμένα παραδείγματα αυτού του συνδυασμού που επιδιώκεται ε, το 2016 και εμεί θα δουλέψουμε σκληρά για να δούμε το πώς θα ε, κάνουμε κάποιες κινήσεις που θα είναι παράδειγμα προς μίμηση και ο σκοπούμενος συνδυασμός είναι αυτό που προωθούμε και έχουμε και κάποια μοντέλα τα οποία εξεργαζόμαστε και έχουμε κάποια χρηματοδοτικά μέσα που ε, συνδυάζουν τα, τον κόμβο παιδικών συμβουλών με την ε, ανάπτυξη, με, την, με τα διαρθωτικά ταμεία πρώτα-πρώτα έχουμε και σε περιφερειακό επίπεδο ε, ενεργήσει και θα συνεχίσουμε. Κατά τρίτο λόγο, ο κόμβος επενδυτικών συμβουλών πρόκειται να συνεργαστεί με τις εθνικές ανεπτυξιακές τράπεζες. Ήδη έχουμε 18 τέτοιες ε, τράπεζες οι οποίες έχουν συμφωνήσει να υπάρξουν κάποια δίκτυα από κοινού τον κόμβο ανταλλαγή καλύτερων πρακτικών, και να μπορούμε να συνεργαστούμε και με τους κατατόπους ε, εμπλεκόμενους στην υλοποίηση των επενδύσεων και των έργων. Και όπως αναφέρετε και εσείς, θέλουμε να δούμε τι θα γίνει στην μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση του πολιετούς πλαισίου και έτσι να διευκολυνθεί ο συνδυασμός των διαρτικών ταμείων με το έτσι. Επίσης να αναβαθμίσουμε το πόσο και πόσους θα καλύψει. Σε συνεργασία πάντα με τον κόμβο συμβουλών. Επίσης ε, τονίζουμε ότι συμφωνεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το να έχουμε πολλά έργα διασυνοριακά θα αποτελέσει προσθεμένη αξία και αυτό και θα ε, ενθαρρύνουμε για την προσθετικότητα και συμπληρωματικότητα είπαμε ότι είναι βασικό χαρακτηριστικό ε, του Ταμείου Στατικών Επενδύσεων και σύμφωνα με το σχετικό κανονισμό τα έργα τα οποία ε, αφορούν την ΕΤΕ, δηλαδή αφορούν τις ε, πιο δύσκολες πτυχές της πολιτικής της έτσι θα θεωρηθούν ότι αποτελούν πρόσθετα στοιχεία. Έχουμε τώρα κάποια νέα ε, προϊόντα τα οποία πρόκειται να καλύψουν και περιφερειακά και τοπικά Ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιες επικρίσεις όσον αφορά την προσθετικότητα και συμφωνούμε ότι η ΕΤΕ πρέπει να προσπαθήσει περισσότερο. Επίσης, τα θέματα της προσθετικότητας πρέπει να καλυφθούν από το σκοπούμενο νομοθέτημα. Επίσης, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την διαφάνεια και αυτά θα πρέπει το νέο νομοθέτημα να καλύψει. Εν κατακλείδη σας τονίζω ότι μόλις ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο το Ταμείο Επενδύσεων και νομίζω ότι ήδη αναμφίβολα θεωρείται πετυχημένο. Άρα, σε σχέση και με το πλάνο Juncker, θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Πρέπει να συνεχίσουμε το έργο μας, ούτως ώστε να έχουμε επενδύσεις στο επίπεδο που θέλουμε. Σας ευχαριστώ και πάλι για τη θετική σας ε, στάση. Είναι σημαντικό αυτό το θέμα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ και για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μπρέσο, έχετε το λόγο πάλι αν θέλετε να απαντήσετε κάποιες ερωτήσεις ή κάποια σχόλια των μελών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σίγουρα δεν είναι δυνατόν τώρα να σχολιάσω εξαντλητικά τα όσα αναφέρθηκα. Μπορώ μόνο να απαντήσω αλλά βέβαια έχουμε τις τροπολογίες, να τα πούμε επ' αυτής της βάσης με τους ε, σκιώδεις εισηγητές για κάποια σημεία. Πάντα έτσι γίνεται όσον αφορά την πρώτη εκδοχή μιας γνωμοδότησης. Νομίζω ότι περισσότερες δυνατότητες δίνονται πέραν πρώτη συζήτηση στη συζήτηση για τις τροπολογίες. Πολύ ενδιαφέρουσα ήταν η συζήτηση ανέκυψαν κάποιες παρατηρήσεις. Ακούσαμε και τις απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και έτσι φάνηκε τι γίνεται με αυτά τα θέματα τα οποία αναφέραμε στην πρώτη έκθεση, όπως θα θυμάστε κύριε το δικό σας κείμενο και είναι κάποια θέματα τα οποία τα αναφέραμε. Και έτσι πρόκειψαν τα σχόλια για την έκθεση της πρώτης χρονιάς. Μα είναι ουσιαστικές αυτές οι απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από αυτών των σχολείων. Και εμείς προσέχουμε πολύ πώς γίνεται η εφαρμογή και η υλοποίηση του Ταμείου. θα πρέπει όλα αυτά τα οποία ζητούμε να ληφθούν υπόψη. Θα πρέπει να έχουμε καλύτερη γεωγραφική κατανομή στα έργα. Θα πρέπει επίσης να υπάρξει περισσότερη ε, ένταξη του ΕΦΣΕ στα διαφορετικά ταμεία ή τέλος πάντων συνεργασία, συνέργεια. Ακριβώς τα ταμεία αυτά να αξιοποιηθούν περισσότερο και να ε, έχουμε επομένως κάποια γενικότερη εφαρμογή και για κάποια έργα υψηλού κινδύνου και επομένως να έχουμε περισσότερο αποτέλεσμα από τις επενδύσεις. Α, το είπε και ο κύριος Μποσινάρο όσον αφορά την προέλευση των πόρων του Ταμείου. Θα πρέπει επομένως να βοηθήσουμε να τρέξουν κάποια έργα και θα πρέπει να κατευθυνθούν αυτοί οι πόροι σε συγκεκριμένες περιφέρειες όπως ακριβώς και το Connecting Europe. Αν αλευθεί υπόψη αυτό, το ειδαφικό στοιχείο και η συνέργεια των επιμέρους πολιτικών των επενδυτικών. Αυτό το αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όπως είπαν και οι συνάδελφοι θα να προσέξουν τι θα γίνει με τον νέο κανονισμό. Ότι δηλαδή αυτό το οποίο θέλουμε θα πρέπει να τα καλύψει ο νέος κανονισμός. Ίσως θα πρέπει να κάνουμε μια ακρόαση, θα πρέπει να συνεργαστούμε με την Επιτροπή των Περιφερειών έτσι και να δούμε πώς θα μπλακούν περισσότερο οι περιφερειακές αρχές και να μην ξεχνούμε ότι εκεί δρούν τα διευθυντικά ταμεία σχεδόν παντού. Και έχουμε τις εθνικές ε, πλατφόρμες που πρέπει εκεί να συμμετάσχουν ε, οι περιφερειακές αρχές έτσι να υπάρξει συνέργεια των ταμείων. Να αξιοποιήσουμε περισσότερο αυτές τις αρχές, τοπικές και περιφερειακές, να ξέρει ο κόσμος τι προβλέπεται, τι προσφέρεται. Όλοι όσοι συναντούμε τις περιφερειακές τοπικές αρχές ξέρουμε ότι και έχονται ενδιαφέρονται για το ταμείο. Αλλά πολλές φορές δεν ξέρουν πώς να κινηθούν. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα πρέπει να συνεργαστεί με αυτές τις πλατφόρμες, με τις εθνικές τράπεζες τελικά, τις ε, επενδυτικές. Να αξιοποιούνται οι πόροι με συνέργειες Και μεγάλο ενδιαφέρον. Ακούσαμε τις προθέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δεύτερη φάση αυτού του, ε, τη, της δεύτερης φάσης λειτουργίας του Ταμείου Επενδύσεων. Καλά, έχουμε τα σχετικά στοιχεία, τα στοιχεία, στοιχεία, αλλά θα πρέπει ε, στα πλαίσια τα οποία υπάρχουν να πετύχει το Ταμείο Επενδύσεων. Μιλάμε για δισεκατομμύρια επενδύσεων. Επενδύσεις που ήδη έχουν ξεκινήσει και έτσι να αποσπάσουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αν θέλουμε να υπάρξει πρόοδος, τότε θα πρέπει να επιτελεστεί ένα έργο το οποίο θα ωφελήσει το σύνολο της Ευρώπης με αυτές τις νέες ευκαιρίες. Και αυτά τα χρήματα να δημιουργήσουν συνοχή. Μια που είναι βασικός στόχος αυτός της πολιτικής της συνοχής. Υπάρχουν πολλές ανάγκες. Αλλά μπορούν να συγκλίνουν οι ενεργειές μας προς το να υπάρξει ομοιογενής ανάπτυξη. Να μην υπάρχουν ασυμμετρίες. Να μην χειροτερέψουν οι διαφορές. Μην γίνουν μεγάλες διαφορές μεταξύ περιφερειών. Άρα θα τα συζητήσουμε αυτά με αφορμή της τροπολογίας και θα προετοιμαστούμε για την επόμενη φάση. Όλα αυτά με ανείχνευση, αναγνώριση της ε, κατάστασης και να δούμε τι κάνουν και οι αρχές που διαχειρίζονται αυτά τα έργα. Να δούμε πώς μπορούμε να τροποποιήσουμε την νομοθεσία και έτσι να υπάρξει πλήρη αξιοπίστη να προφύγουν όσο γίνεται αυτή η πόρη. και με τέτοιο τρόπο που να κατατείνουν στην επίτευξη των στόχων δηλαδή την περιφερειακή και γενικότερη συνοχή αυτά που είναι σημαντικοί στόχοι μας Σας ευχαριστώ πολύ Ολοκληρώνεται εδώ η συνεδρίαση για σήμερα το πρωί, αφού ολοκληρώσαμε και το θέμα αυτό. Μπορούμε να συνεχίσουμε αμέσως με τη συνεδρίαση των συντονιστών. Γι' αυτό λοιπόν οι συνάδελφοι οι οποίοι δεν συμμετέχουν σε αυτή τη συνεδρίαση παρακαλώ να αποχωρήσουν από την αίθουσα.